Good afternoon, everybody. Good afternoon, colleagues. As our... Uh, Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Επειδή ο πρόεδρος μας λείπει σήμερα, θα προεδρεύσω εγώ στην απόψινή συνεδρίαση. Έχουμε κάποιους ε, σημαντικούς προσκεκλημένους ε, απόψε. Θα, ακούσουμε, ε, θα τους ακούσουμε και θα τους θέσουμε ερωτήσεις. Καταρχήν ε, θα υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας πω ότι το σημείο 6 που αφορά τις απαιτούμενες βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στα έγγραφα κατόπιν της θέσης ισχύ της Σύνθηκης της Λισαβόνας ακυρώνεται ναι. λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του εισηγητή. Οι πολιτικές ομάδες θα αποφασίσουν αν θα υποβάλουν τροπολογίες Ε, οπότε θα επανεξετάσουμε το θέμα. Σε σχέση με το σημείο 5, η νομική υπηρεσία του ΕΛΚ, ε, του Ευρωπαϊκού μάλλον Κοινοβουλίου, θα μα κάνει μια παρουσίαση πριν από την ψηφοφορία. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσει για την ημερησία διάταξη, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Ωραία, λοιπόν. Μετά έχω να σα κάνω και μια ανακοίνωση σε σχέση με τον ορισμό των εισηγητών. Οι συντονιστέ μα ε, συστήνουν να ορίσουμε τον εισηγητή για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την τήσια έκθεση δηλαδή για τα δικαιώματα στην Ένωση και ο ε, μένα όρισαν ως εισηγήτρια ή συντονιστές. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι γίνεται δεκτή η πρόταση. Και τώρα τα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη, συμπεράσματα και επανεξέταση της Σουηδική Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Έχουμε παρουσίαση από την κυρία Μπέατρι Άσκ, τη Σουηδή Υπουργό Δικαιοσύνη. Πείτε μας λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ε, πώς, ε, ποια είναι η άποψή σας για τα επιτεύγματα της Σουηδικής Προεδρίας και αναφέρομαι βέβαια και στο μακροσκελές έγγραφο το που αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η κυρία Άσκα είναι υπεύθυνη για τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά δικαιώματα, τα, τα εσωτερικά συγγνώμη, ε, άρα λοιπόν είναι υπεύθυνη αρμόδια για αυτό το θέμα. Αν έχετε ερωτήσεις παρακαλώ να περιμένετε γιατί αργότερα στις 4 θα έχουμε και την... τον Υπουργό Τομπία Μπίλστρομ για τα θέματα μετανάστευση και ασύλου. Κυρία Άσκη, σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε για την ε, συνεργασία σας μαζί μας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Περίπου τρει μήνε έχουν περάσει από την τελευταία μου παρουσία εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να σα παρουσιάσω τι προτεραιότητε και φιλοδοξίε τη Σουηδική προεδρία. Έκτοτε έχουν γίνει πολλέ έντονε προσπάθειε καθώ και έντονη συζήτηση κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και νομίζω πω πλέον είναι και η ώρα για να σα αναφέρω τα όσα πετύχαμε στον τομέα τη δικαιοσύνη και των ιστορικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια της Προεδρία. Προεδρίας. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι τα θέματα αυτά ήταν μεγάλης προτεραιότητα στην ατζέντα μας και προσπαθήσαμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας αλλά και για την προστασία της ε, κεραιότητας των ε, πολιτών μας. Οι πολίτες ήταν στο επίκεντρο της εργασίας μας, θέματα όπως ε, διαδικαστικά δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων ήταν πολύ σημαντικά. Η προοπτική του πολίτη επίση ήταν ξεκάθαρη όταν εργαστήκαμε επί του προγράμματος της Οκχόλμης, το οποίο βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής καθώς και στι απόψει των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κοινωνία των Πολιτών, των διαφόρων ευρωπαϊκών σωμάτων και επίσης βασίζεται στις εντατικέ έντονε συζητήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη που τη συναποτελούν. Εγώ μαζί με τον Τομπία Σεμπίλστρομ συμμετείχαμε στην σύνταξη του προγράμματο τη Στοκόλμη που έγινε στο, μια συνεδρίαση που έγινε στο Στρασβούργο στι 24 Οκτωβρίου. Το περιεχόμενο του ψηφίσματος ολοκληρώθηκε μετά από τη σημαντική συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο. Στη... Επίσης το συζητήσαμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και συμφωνήσαμε τη αρχή για, το ουσιαστικό για την ουσία του. Αυτό που τώρα μας μένει είναι η εξέταση από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που και ελπίζουμε να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 10 και 11 Δεκεμβρίου ανοιχτή Ευρώπη όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του ατόμου. Η προοπτική του πολίτη θα πρέπει να, να χρησιμοποιηθεί ως σημείο κίνησης για, για την εργασία μας. Επίσης, η συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ακαιρεότητα των δικαιωμάτων του ατόμου, του ανθρώπου το... Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Εκχόλμης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιδέα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνυπογράψει στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών όσο γίνεται πιο σύντομα. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να γίνουν όλα αυτά, να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο σύντομα και υπολογίζουμε, στην, βασιζόμαστε και στη δική σας ε, βοήθεια και υποστήριξη. Όσον αφορά το διασυναρικό έγκλημα, η πρόκληση είναι ε, πολύ μεγάλη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα διοικητικά σύνορα να εμποδίζουν τα όργανα πρόληψης του εγκλήματος να διεξάγουν το έργο τους. Χρειάζεται κοινέ λύσεις για τα κοινά προβλήματα. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αυτό το τομνίζει ώστε να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου προβλήματα. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό η ανταλλαγή πληροφοριών και τα βασικές προδιαγραφές για την προστασία της ε, ιδιωτική ζωή των ανθρώπων να συγκεντρώνονται αλλά να μην αποθηκεύονται περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Θέλουμε να έχουμε μια ασφαλή Ευρώπη που το διασυνοριακό έγκλημα θα κατοπολεμάται αποτελεσματικά ενώ θα γίνεται σεβαστή η προσωπική ακαιρεότητα. Η αρχή της αμοιβέ αναγνώρισης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εξυπηρετεί ως θεμελιώδης αρχή της συνεργασίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκτελούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα δικαστήρια άλλων χωρών και χρειάζεται για κάτι τέτοιο αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ένας τρόπος για την αύξηση αυτής της εμπιστοσύνης είναι το να αυξηθεί η γνώση σχετικά με τα δικαστικά συστήματα της κάθε χώρας. Ε, περιλαμβάνονται εδώ προτάσεις για την τα βελτιωμένα εκπαιδευτικά μέτρα, ε, προγράμματα ανταλλαγών εισαγγελέων και δικαστών, καθώς και η διεύρυνση των υφιστάμενων δικτύων. Επίσης, τα ελάχιστα κοινά δικαιώματα για την υπεράσπιση των ε, κατηγορουμένων, όπως η μετάφραση και στο πρόγραμμα υπάρχουν βήματα για τη βελτίωση των διαδικαστικών δικαιωμάτων. Εκείνοι που είναι θύματα εγκλημάτων επίσης ε, λαμβάνονται υπόψη όλος ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης όπου υπάρχει σαφής προοπτική ε, για τα θύματα των εγκλημάτων και αυτό είναι νέο στοιχείο η Σουηδική Προεδρία έχει κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε ε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης να ανταποκριθεί στις επιθυμίες των πολιτών. Θέλουμε ένα φιλόδοξο και συγκεκριμένο πρόγραμμα με σαφείς προτεραιότητες και πιστεύω πως όντως το πετυχαίνουμε. Τώρα προσβλέπουμε στην υιοθέτηση του προγράμματος της Στοκχόλμης ε, στο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου έπειτα θα εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επερχόμενη Σουηδική Προεδρία να φτιάξουν ένα πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος Στοκχόλμης. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό έργο και προσβλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επικοδομητική συνεργασία. Αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, πέρα από το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη, η Σουηδική Προεδρία έχει εργαστεί με διάφορα άλλα θέματα ε, και μέσα. Α πούμε, επαναλήφθηκαν οι συζητήσει για τα δικαιώματα τα διαδικαστικά κατά τη διάρκεια δικονομικά κατά τη διάρκεια των ε, ε, των ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με αυτή, μέσα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, ένα σημαντικός εταίρος στην καταπολέμηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων, η Σουηδική Προεδρία έχει εστιάσει την προσοχή στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης και ένα συγκεκριμένο έγγραφο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο την 1η Δεκεμβρίου και αυτό θα χρησιμεύσει ως κατευθυντήρη γραμμή για την εργασία μας σε αυτό το τομέα. Εκεί εμπετεύχθη ευρεία συνένεση όσον αφορά τις ευρείε γραμμές για τις διαπραγματεύσει για την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων, αυστηρότερες ποινές και καλύτερη προστασία των θυμάτων εγκλημάτων. Με την έναρξη ισχύω της, της συνθήκης της αναμένουμε αυτή η συμφωνία να αποτελέσει τη βάση για μια οδηγία για τα ε, εμπορία των, ανθρωπων... των ανθρωπίνων όντων, των ανθρώπων ε, και αυτό θα συμφωνηθεί μαζί με το Κοινοβούλιο μέσα στη διαδικασία της συναπόφαση. Η καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρωπίνων όντων απαιτεί κοινά μέσα. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές που είναι πολύ προσιλωμένοι σε αυτά τα θέματα, το πώς δηλαδή θα καταπολεμηθεί η εμπορία των ανθρωπίνων όντων. Άλλη μια προτεραιότητα της ειδική Παιδείας ήταν η καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και της ε, ε, σεξουαλικής κατάχρησης. Και εδώ χρειαζόμαστε σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ενός καλύτερου νομικού πλαισίου και ελπίζουμε πως θα είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε σχετική οδηγία στην ε, διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Ξεκινήσαμε επίση μια εθελοντική οικονομική συνεργασία για να καταπολεμηθεί η παιδική πορνογραφία στο ίντερνετ. Σημαίνει συνεργασία μεταξύ τραπεζών, ε, εκκλησιών, τραπεζών ε, για να μπορούν να σταματήσουν τη χρηματοδότηση της ε, παιδικής πορνογραφίας και αυτό συμφωνήθηκε σε υπουργική διάσκεψη τον Οκτώβριο. Καλύτερα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε δε τα εγκλήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βελτιώνονται οι επικοινωνίες, καθώς ε, ε, η σύγχρονη τεχνολογία αναπτύσσεται, γίνεται και πιο εύκολο η πιο εύκολη μετάβαση των εγκληματιών από μια χώρα στην άλλη. Είναι λοιπόν κοινή μας ευθύνη να καταστήσουμε ευκολότερη την ε, σύλληψή τους από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους. Και η συνεργασία μεταξύ αυτών των αρχών είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια γενική συνολική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, γιατί ο στόχος είναι να έχουμε ε, μια αποτελεσματική διαχείριση που θα οδηγεί στην επιτυχή και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών. Σημαίνει επίσης ε, συγκεκριμένους όρου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη ιδιωτική ζωής. Ε, διαπραγματευτήκαμε και μια προσωρινή συμφωνία με τις ΕΠΑ για την πρόσβαση στις πληροφορίες από το SWIFT. 13 Νοεμβρίου έγινε δεκτή αυτή η συμφωνία από το Συμβούλιο των Υπουργών. Προσπαθούμε επίσης να αποφύγουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Άλλη διεθνής υποχρέωση. Χρειάζεται να συνεργαστούμε σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης για να καταπολεμήσουμε το, την τρομοκρατία. Και Διαπραγματευτήκαμε συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης ε, με τη ΣΥΠΑ μέσω του SWIFT και ελπίζουμε πως ε, την επόμενη χρονιά θα καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης για κάποια πιο μόνιμη απόφαση σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Συνδική Προεδρία επίσης έχει επιλέξει να αγωνιστεί για την ποιοτική ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συμφωνήσει για μια, οδηγία για την ε, αδειοδότηση λειτουργίας των ιατροδικαστικών εργαστηρίων, ούτως ώστε να έχουμε υψηλά επίπεδα ε, και προδιαγραφές πράγμα το οποίο υιοθετήθηκε για την ε, δημιουργία ενός ομοιόμορφου συστήματος ε, για την ιατροδικαστική ανείχνευση ναρκωτικών και αυτό για την καταπολέμηση της χρήσης και κατάχρησης ναρκωτικών στην Ένωση. Έχουμε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ε, παραγωγή κοινή νομοθεσία όσον αφορά την καταπολέμηση των εγκλημάτων. Όμω, προαπαιτούμενο για κάτι τέτοιο σημαίνει αύξηση τη εμπιστοσύνη ανάμεσα στι αρμόδιε ε, αρχέ θα πρέπει να μπορούν να συνομιλούν άμεσα μεταξύ του. Στο πλαίσιο του προγράμματο Στοκχόλμη θέλουμε να θεσπίσουμε φιλόδοξου στόχου για την κατάρτιση των αξιωματικών, των εισαγγελέων και των δικαστών, συμπεριλαμβανομένη ανταλλαγή ε, όλων αυτών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, τον Οκτώβριο καταφέραμε να διοργανώσουμε μια άτυπη υπουργική συνεδρίαση στη Χάγη για να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα αυτό. Και με την ε, έναρξη ισχύω τη συναπόφαση για τη Europol, είμαι συμπεπισμένη ότι η σημασία αυτού του οργανισμού θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυξάνεται και η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών ε, σε ολόκληρη την Ένεση. Άλλη σημαντική, άλλο σημαντικό τομέα είναι οι εξωτερικέ ε, σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και τη δικαιοσύνη. Τον φθινόπωρο είχαμε σχετική υπουργική συνάντηση με του στρατηγικού μα εταίρου, με τη ΣΥΠΑ, δηλαδή τη Ρωσία και με τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Στην υπουργική διάσκεψη με τη ΣΥΠΑ Υιοθετήθηκε από κοινού η δήλωση της Washington που θεσπίζει το πλαίσιο για την διαδροτική συνεργασία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, η ΕΕ και η ΕΠΑ συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία ώστε να καταπολεμήσουν τα σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα, δηλαδή ε, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, ε, εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο ανθρωπίνων όντων, καθώς και προστασία ατομικών δικαιωμάτων. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που πετέφθησαν από την Προεδρία από το φθινόπωρο. Ήταν πολύ εντατική η εργασία μας συναρπαστική. Πολλές προσπάθειες καταβλήθηκαν από εμά, από την Κομισιόν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω πως τα, όσα καταφέραμε και τα μέτρα που υιοθετήσαμε από κοινού κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας θα οδηγήσουν σε μια πιο ανοιχτή και πιο ασφαλή Ευρώπη για εμά και τους συμπολίτε μας. Εύχομαι λοιπόν πως οι συμπολίτε μας θα ανακαλύψουν και θα μπορέσουν να καταλάβουν πόσο πολύ σκληρά εργαστήκαμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια ευχαριστεί την Υπουργό. Δεν έχει ανοίξει το μικροφωνό της η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε και το έργο που επιτελέσατε. Uh, Ένα σωρό συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μπουσούτιλ πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για την εισήγησή σας ε, θα ήθελα να λάβω το λόγο για να σας ευχαριστήσω για το έργο το οποίο επιτελέσατε κατά την Προεδρία αυτού του εξαμήνου και Νομίζω ότι καθώ μια φορά ε, έχετε δύο βασικά επιτέματα. Πρώτα από το πρόγραμμα τη Στοχόλμη και δεύτερον τη θέσπιση, τέλο πάντων τη θέση ισχύ τη νέα συνθήκη. Με το οποίο θέμα και ξεκινώ, όπω γνωρίζετε, ε, θεωρούμε ότι τώρα μπορούμε να ανατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα, θετικά και δυναμικά. Τώρα μια που θα τεθεί σε ισχύ αυτή η συνθήκη η οποία ε, θα μας κάνει να έχουμε λέγεν σε έναν τομέα όπου θα είναι μεγάλη διαφορά για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη και καθημερινή του ζωή. Όπως είπατε, το θέμα της δικαιοσύνης είναι πραγματικό και καίει τους πολίτες. Επομένως, θα κάνουμε εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο ε, θα, θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί. Γιατί ε, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα ανακύψουν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, δηλαδή το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε την Σουηδική Προεδρία διότι το θέμα το προώθησε, το διεκπαιρέωσε και όπου να είναι θα γίνει τις επόμενες μέρες η οριστική έγκριση. Νομίζω όμως ότι προλιάνατε το έδαφος για κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί, μια που εσείς είχατε την Προεδρία τώρα ε, που ήρθε η ώρα για αυτό το θέμα, οπότε και αυτόν τον τρόπο ε, είχατε ατού στα χέρια σας και το εκμεταλλευθήκατε όπως έπρεπε. Από ε, την άλλη μεριά, αυτό το οποίο μας απασχολεί δεν είναι μόνο αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο πρόγραμμα της Στοχόλμης και θα πρέπει να προσθέσω ότι ακόμα δεν έχει πέσει στα χέρια μου η οριστική μορφή του προγράμματος που σήμερα μόλις ολοκληρώθηκε όμως έχω δει κάποιες ε, προηγούμενες ε, εκδόσεις, ίσως μπορείτε εσείς να μας διαφωτίσετε λίγο πάνω σε αυτό και ε, το, το, το, αυτό που έχει σημασία είναι το πρόγραμμα της Στοχόλμης και το πώς θα μπορέσουμε αυτό να το υλοποιήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για μας, ιδίως εδώ στην, στο, στο Κοινοβούλιο, στη δική μας πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ. Επομένως, με μεγάλη προσοχή θα παρακολουθήσουμε αυτό το ζήτημα της ε, ε, εφαρμογής. Τώρα, για τα θύματα των τέτοιων εγκλημάτων, τα δικαιώματά τους, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, εμείς πρόκειται να αναλάβουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως επίσης και το θέμα των δικαιωμάτων των ανηλίκων, στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε και επίσης θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσει η Ευρώπη να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αφήσατε κληρονομιά και την οποία θα πρέπει υπάρξει να την συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις μαζί, θέλετε να απαντήσετε τώρα. Ό,τι θέλετε, λέει η κυρία Υπουργό. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι άλλες ερωτήσεις έχουμε. Οι μπορεί να κολλάνε. Γιατί αφορούν τα ίδια θέματα. Άρα θα είναι πιο εύκολο. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag die over ditzelfde onderwerp gaat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 van eh, personen en entiteiten. Θα ήθελα να αναφερθώ στις, στους περιορισμούς ε, σχετικά με που επιβάλλονται σε άτομα που εμπλέκονται στα δίκτυα της Αρκάιντα, του Μπιν Λάντεν κτλ. Είχαμε καταλάβει από όσα είχε πει η Σουηδική Προεδρία ότι το Συμβούλιο επρόκειτο στη συνεδρία της 30 Νοεμβρίου να εγκρίνει τις θέσεις του. Γιατί. Γιατί το θέμα αυτό δεν περιελήφθη στην ημερήσια διάταξη της 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται να καλυφθεί ε, το θέμα υπό όρους της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερως γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να μάθω και γιατί αυτή η αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ κυρία Χένης Πιώσετ και μετά θα σας δώσω το λόγο κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. περίμενα και εγώ να ακούσω την απάντηση στην ερώτηση γιατί εγώ την, την κατάλαβα καλά παρότι είναι στη δική μου γλώσσα. Ε, δεν θα επαναλάβω τα εγκομιαστικά λόγια του κυρίου Μπουσούτη ωστόσο οφείλω και εγώ να πω ότι με μεγάλη χαρά σας βλέπουμε εδώ ε, από την καρέκλα της Προεδρίας. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και εγώ για το SWIFT. Ανάμεσα στο signing και το concluding, δηλαδή την υπογραφή και τη σύναψη μιας συμφωνίας, υπάρχει προφανώς διαφορά. Αυτό δεν με εκπλήσει, έστω. Αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί επελέγει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει τις θέσεις του. Γιατί μην μου πείτε ότι εξ αρχής μας είχε προειδοποιήσει το Συμβούλιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά, και εξεπλάγημεν όταν ε, μάθαμε ότι για τη μεταβατική αυτή έκθεση ε, θα είχαμε και εμείς λόγο. Γιατί λοιπόν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πώς ξαφνικά εδόθη στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα της παρέμβασης στη διαδικασία. Για το SWIFT, η ιδέα της αμοιβαιότητας για την οποία ε, διαρκώς γίνεται λόγος ως προς τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, όσο η όσο η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικό της σύστημα, το δικό της πρόγραμμα, ε, δεν μπορούμε να είμαστε απαιτητικοί. Και μάλιστα από την Επιτροπή μας είχαν απαντήσει ότι το κόστος ήταν πολύ ψηλό και μικρό το όφελος. Εσείς σε αυτό τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Άσκ, παρακαλώ να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις και μετά θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά με την οποία τυπώθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό να ε, έχουμε ένα πρόγραμμα ως Προεδρία και να το ακολουθούμε με τη σειρά, μία προεδρία μετά την άλλη. Υπάρχει, ένα πρόγραμμα για το... Υπάρχει το πρόγραμμα Στοκχόλμης, το οποίο θα συνεχίσει μετά με τη σειρά της να εφαρμόζει και η Ισπανική Προεδρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το σχέδιο αυτό εφαρμογής να τηρηθεί, γιατί πολύ συγκεκριμένα μέτρα θα προβλεφθούν με βάση και τις φιλοδοξίες που προτείνει το ε, πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Από την ε, προηγούμενη Παρασκευή βλέπουμε ότι διαρκώς ε, εκφράζονται ε, εκφράζεται η ανάγκη για ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδιαίτερα της εγκληματικότητας βάρος των παιδιών. Και εμείς βεβαίως θέλουμε οι δικαστικές μας αρχές να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις πτυχές ε, της εγκληματικότητας που στρέφεται κατά των παιδιών. Για την κυρία Βόσκουρτ, για τους περιορισμούς και την ε, καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Είναι ένα ζήτημα, εξ γνωρίζω, το οποίο αφήνεται των αρμοδιοτήτων των Υπουργών Εξωτερικών και όχι των Υπουργών Εσωτερικών. Στη δική μας μέρη διάταξη δεν υπήρχε το θέμα αυτό. Άρα δεν μπορώ να είμαι σε θέση να απαντήσω. Άλλωστε μου φαίνεται κάπως ε, παράξενο να, να υπήρχε πιθανότητα να συζητηθεί στο δικό μας επίπεδο, γιατί θα ήταν θέμα μάλλον των Υπουργών των Εξωτερικών. Για δε το SWIFT και γιατί προβλέφθηκε το χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε. Να σας πω. Είχαμε την ανησυχία ότι μπορεί να ε, η ανταλλαγή απόψεων, να μην είναι παρκής και φοβηθήκαμε ότι μπορεί κάποια σημεία να μην καλύπτονται. Και έτσι θελήσαμε τις πληροφορίες να τις καλύψουμε βάσει και τα στοιχεία που έχουμε για το αμερικανικό σύστημα για να λειτουργεί το σύστημα με βάση τους κανόνες. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το επιδιωκόμενο για μας αποτέλεσμα και από την άλλη βέβαια έχουμε απόλυτη συνείδηση του περίπλοκου του συστήματος. Έχουμε συζητήσει, κάναμε τις διαπραγματεύσεις μας και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμη ε, συζητήσει το θέμα αυτό. Επανειλημμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθαμε για να συζητήσουμε και τα θέματα αυτά, αλλά ε, πάνω απ' όλα θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε να ξέρουμε, και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας απαντήσω προς το χρονοδιάγραμμα, ότι δεν, θέλουμε, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή οι ελλείψεις ως προς την παρακολούθηση του συστήματος SWIFT. Γιατί δεν έχουμε κανένα περιθώριο να αφήσουμε ακάλυπτες τις κινήσεις κονδυλίων των τρομοκρατών, πόρων των τρομοκρατών. Αυτό ήταν κάτι το οποίο συζητήσαμε από πριν και Είσαστε ήδη ενήμεροι. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ακούσαμε τρεις ε, συναδέλφους, ακούσουμε άλλου τρει Και μετά μπορείτε πάλι να λάβετε το λόγο και εσεί για να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Άλμπρεχτ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με χαρά βλέπω ότι έγιναν δεκτές κάποιες από τις παρατηρήσεις μας στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης σε θέματα του εσωτερικού και της δικαιοσύνη, ιδιαίτερα προς την <laughs> προστασία των προσωπικών δεδομένων, που μας ενδιαφέραν μας ιδιαίτερα. Και βλέπω ότι ε, ναι μεν έχουν συμφωνηθεί πράγματα θετικά πράγματα ικανοποιητικά, αλλά τα πάντα θα κρυθούν από την υλοποίηση. Γι' αυτό θα ήθελα να δω αν υπάρχει άλλη ευκαιρία να ε, συζητήσουμε αυτά τα πράγματα αργότερα και να έχουμε βέβαια και την κατάλληλη ανταλλαγή ε, ε, μέρος πληροφόρηση. Για τη μετανάστευση όμως ε, και τους πρόσφυγες υπάρχουν άλλα θέματα στα οποία δεν είμαστε και τόσο ευχαριστημένοι, το οποίο θα έπρεπε να θίξουμε. Ε, στο SWIFT επίσης, το οποίο εθίγει νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω σε, αυτή την, ε, σε αυτό το θέμα να γίνει η συζήτηση ανοιχτά και με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ότι όταν έχουμε λάβει, όποτε λάβαμε την ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όποτε μπορέσαμε να σχηματίσουμε την εικόνα της κατάστασης εμείς ως Κοινοβούλιο, μπορούμε και να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις. Είμαι πεπισμένος ότι το ίδιο θα συμβεί και στην υπόθεση του SWIFT. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι πολλά γίνονται και κλεισμένων των θυρών, επικρατεί μια, ε, ένα πέπλο μυστηρίου και σιωπής ενώ θα ήθελα να ε, ακούσω από πλευρά σας κάποια υπόσχεση ότι το Κοινοβούλιο, δυνάμει της Συνθήκης Λισαβόνας, θα ενημερωθεί πλήρως, θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις τόσο για το SWIFT όσο και για άλλα θέματα που είχαμε, για τα οποία είχαμε εκφράσει την επιθυμία στο παρελθόν Τώρα βλέπω ότι ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά και θα ήθελα να ακούσω ε, εάν έχει το Συμβούλιο για τα θέματα των ιστορικών και της δικαιοσύνη την πρόθεση να ε, επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία και τη συναπόφαση φυσικά, αλλά και την αξιολόγηση των μέτρων. Ευχαριστώ κύριε Αλπρέχτη, κυρία Ινετφέλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για την ε, συμμετοχή σε εργασίες μας κατά αυτήν την τόσο σημαντική ε, περίοδο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αφαιρθώ σε διάφορες ε, διεθνείς συμφωνίες, καταρχάς το SWIFT. Ο λόγος, από ό,τι έμαθα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, για τον οποίο τώρα προχωρεί η διαδικασία με τη σύμφωνη γνώμη ήταν ότι οι τέσσερις χώρες επικαλέστηκαν το άρθρο 24.5, 24.5 παράγραφος, με την επιφύλαξη λέει, της κοινοβουλευτικής εξέτασης, πράγμα το οποίο δεν επέτρεψε στο Συμβούλιο λύση άλλη από αυτήν της ε, σύμφωνης γνώμης. Πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να είχαμε ενημερωθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα ακόμη είχαμε τη συζήτηση και δεν μας είπε κανείς τίποτα. Επίση, είπατε μόνοι σα ότι θα πρέπει επικόντω να εγκριθεί η νέα συμφωνία SWIFT. Αλλά θα υπενθυμίσω ότι το 2007 ήδη γνωρίζαμε, πριν από δύο μισή χρόνια ε, γνωρίζαμε ότι θα άλλαζε ριζικά η δομή η αρχιτεκτονική του προγράμματος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα. Αλλά έστω. Επίση, μα λέτε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει χάσμα στην μεταφορά δεδομένων. Πολύ καλά, να σας πιστέψω σε αυτό αλλά μια θα σύμφωνη μας γνώμη. Δεν θα πρέπει αυτές τις πληροφορίες να μας τις γνωστοποιήσετε. Διαφορετικά, πώς θα λάβουμε την απόφαση, επί την βάση. Και άλλη μία πιο γενική ερώτηση που αφορά τις ε, διεθνείς συμφωνίες. Τι χρονοδιάγραμμα προβλέπετε για, να, ε, για την υποβολή του θέματος προς έγκριση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο μα ε, απασχόλησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να προχωρούμε ταχύτατα. Η Επιτροπή όμω, η οποία καλύτερα να καταθέσει τι προτάσει προ το Συμβούλιο, φαίνεται να θέλει να καθυστερήσει όλη τη διαδικασία μέχρι τον Ιανουάριο. Και να αρχίσει μόνο τότε. Το Συμβούλιο τι θέση έχει γι' αυτό. Γιατί φυσικά αυτό το ερώτημα έχει να κάνει και με το SWIFT και με δύο άλλες ε, διεθνείς ε, συμφωνίες, αλλά και γενικότερα με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Χωρίς να υπάρχουν λοιπόν προθεσμίες στην ε, συνθήκη, η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης μπορεί να δίνει στο Κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει νόημα μόνο εφόσον το Κοινοβούλιο είναι ενήμερο εγκαίρος. Μάλιστα δεδομένου ότι κάποια έγγραφα κυκλοφορούν δίπλα στο φωτοτυπικό και τα βλέπουμε τυχαία, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες προτάσεις για έγκριση ειδικών ρητρών στις οποίες έχει αντιταχθεί το Κοινοβούλιο ε, επί μεγάλο διάστημα. Και πάλι με τη νέα διαδικασία, όπως συμμετέχει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Φυσικά αυτό ισχύει και για τις συμφωνίες, για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την υπερατατική Συμφωνία. Παρακαλώ λοιπόν να ενημερώσετε το Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό. Η κυρία Μακοβέη. Thank you. Um, I also... Ευχαριστώ. Ναι, κύριε και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Σουηδική Προεδρία για το που και για την συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για το ότι αναφέρεται το πρόγραμμα τη ε, της Στοχόλμης ε, την διαφθορά στην ιδιωτικό τομέα και με την ευκαιρία αυτή να ενημερώσω όλου ότι την Τετάρτη αυτή τη εβδομάδα στι 9 Δεκεμβρίου από τις 10 με 12.30 υπάρχει μια δημοσία εκδήλωση ε, που συνδιοργανώνεται ε, από διάφορους εξημών ε, και με την Transparency International. Μια που αυτή η μέρα είχε αφιερωθεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί το κείμενο το οποίο σήμερα το πρωί λάβαμε έχουν επισημάνω δύο τινά. Πρώτα πρώτα ότι στο 445 445 δηλαδή, εκεί που λέει οικονομικό έγκλημα και διαφθορά, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσουν κάποιους δείκτες για την καταβολέμηση της ε, διαφθοράς και επίσης να εκπονηθεί και μια σχετική πολιτική. Και αυτό να γίνει ε, σε συνεργασία με, το, με την αντίστοιχη επιτροπή, το αντίστοιχο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κυρία Υπουργέ, θα στείλω σχετικά ένα, ένα email. και αυτά τα, τα, τα στο Στρασβούργο και αναφέρεται στην ίσα με την Κυριακή, αυτό το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπη. Συμφωνώ με αυτό βεβαίω. όμως δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποκαταστήσουμε έτσι το, ότι την ανάγκη ύπαρξη δικού μα μηχανισμού για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την διαφθορά. Μόνο θα προκύψει μια προστιθέμενη αξία. Μόνο αν έχουμε αυτό το δικό μας ε, όργανο, το δικό μα φορέα. Έτσι θα βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά σε σχέση με το τι θέλουμε να γίνει από το Συμβουλίο τη Ευρώπη. Στο πρόγραμμα τη Στοκχολμής θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα αναφέρεται ένα σχετικό μηχανισμό που κατά τη γνώμη μου τώρα επιδέχεται ε, περαιτέρω επεξεργασία, διότι δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να λέει κάτι γνώμη μου. Το πώ θα γίνει η εφαρμογή αυτών των αρχών. Ότι χρειάζονται κάποιοι εικονισμοί, χρειάζεται κάποια διαδικασία, ούτως ώστε να παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει στα κράτη-μέλη. Δάλλως θα καταλήξουμε με πάρα πολύ ωραία λόγια που θα διατυπώνουν ε, επί χάρτου μόνο ε, την πολιτική χωρίς να υπάρχει κάποια συνέχεια. Αυτό ήθελα να σας πω, το που με προβληματίζει και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε όλοι όσοι θέλουμε κάτι από όλα αυτά τα λόγια να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, θα δώσουμε κυρία ε, την κυρία Υπουργό, το λόγο για να απαντήσει όλε αυτέ τι ερωτήσει και κατόπιν θα γίνει ένα τελευταίο τελικό γύρο τραπέζι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα και τον κύριο Άλμπρεχτ. Έχω να πω ότι έχει δίκιο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Όμω δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό το οποίο είπατε και μα λέει και σύμφωνο. Διότι το πρόγραμμα τη Κοπεχάγη είναι αρκετά γενικόλογο. Είναι αρκετά σφαιρικό που δεν προβλέπει ε, λεπτομερείς ε, για όλα σχεδόν τα θέματα. Άρα, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι θα πρέπει να διεκπαιρώσουν το θέμα προς την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε. Για το SWIFT έχουμε επεξεργαστεί το θέμα όσο μπορούσαμε και κάναμε ό,τι θεωρήσαμε ότι είναι δυνατόν και θεωρήσαμε ότι το πιο βασικό είναι να υπάρχει ανοιχτή μας στάση. Όμως, υπήρχαν κάποιες περιπλοκές, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες που φαντάζομαι τις γνωρίζετε. Οπότε ακόμα και μια τέτοια άτυπη συμφωνία πρέπει να περάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο ε, εδώ και καιρό το επιδιώκαμε. Και όταν λέμε για ανοιχτή στάση για μας ήταν θέμα κλειδί σε όλη την Προεδρία ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα χαρτιά μας συνεχώς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο θα πρέπει με τη σειρά του να δείξει θετικό πνεύμα, να δείξει επικοδομητικότητα όταν έρχεται η ώρα ε, να, να, να, να κάνει ο καθένας μας από ένα βήμα πίσω και να υπάρξει συμφωνία. Και περιμένω από εσάς επομένως έτσι τέτοια θερμή, στα θερμό ενδιαφέρον. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα άρουμε κάθε κάθε πρόβλημα πώς θα σταματήσουν υπάρχουν στεγανά που εμποδίζουν την ε, πρόοδο του θέματος. Και δεν μιλάω τώρα για καμία συνωμοσία της θεωρίας, ε, γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όμως, πάρα πολύ σκληρά προσπαθούμε, ούτω ώστε να υπάρχει διαφάνεια να είναι όλα ανοιχτά. Να ανοίξουν επομένω αυτέ οι διαδικασίε, να ανοίξουν οι διαπραγματεύσει. Αν δεν υπάρχουν δικοί κανόνε, α δουλέψουμε του κανόνε που έχουμε. Βεβαίω και υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά, βεβαίω και θα ήθελα και εγώ να απαντήσω σε πάρα πολλά ερωτήματα, όμω απαντώ μόνο σε ό,τι μπορώ. Και, και άρα, εμεί θα συνεχίσουμε ε, αυτό τον δρόμο, αυτή την πορεία τη ανοιχτή, τη ελεύθερη συζήτηση που νομίζουμε ότι είναι ο πιο εύκολο, ο πιο σωστό τρόπο για να βρεθούν οι απαντήσει. Όπω σα προείπα, δεν είμαστε μόνοι μα. Πολλοί εμπλέκονται πολλοί που έχουν άλλου είδους παράδοση, όχι τόσο ανοιχτής στάσης. Τώρα, κυρία Νετφέλτ. Ελπίζω ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα καταφέρουμε πριν το τέλος του έτους και φυσικά αφού και εσείς έχετε δώσει ε, την, την, το πράσινο φως. Το πρόβλημα είναι ότι δεν προβλέπονται τίποτε κανόνες σε σχέση με το πώς οφείλουμε να ενεργήσουμε. Επομένως, προσπαθούμε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει, πώς το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να έχει στα χέρια του τα σχετικά έγγραφα, ε, εγκαίρος κλπ. Κύριε Μακοβέση, ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είσαστε η μόνη ε, ευρωβουλευτή που ήρθε να με βρει, που ήρθε σε επαφή μαζί μου μετά αυτή τη συνεδρία του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, είπατε πολλά θέματα, έχετε δίκιο, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα που να κάνουμε και περισσότερα και ε, θα πρέπει σε συνεργασία με το Συμβούλιο να τεθούν κάποια κριτήρια για το τι θα κάνουμε. Έχουμε δύο παράλληλα και θα πρέπει με τη σειρά μας να φροντίσουμε να είναι συγκρίσιμα. Ιδάλλως, θα έχουμε επικαλύψεις. Ελπίζω, όπως βοηθήσατε μέχρι τώρα, να συνεχίσετε να βοηθάτε. υπονομεύσουμε τις αρχές οι οποίε ε, θα μας βοηθήσουν κανονικά να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. σε ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Και τώρα ο τελευταίος γύρος ερωτήσεων με πρώτη την κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν αναφερθώ στο πρόγραμμα της Στοκχόλμη, θα ξεκινήσω με το SWIFT. Δεν έχω υπερβολικές ελπίδες γιατί και από την προηγούμενη εβδομάδα ε, κατάλαβα ότι υπάρχουν ε, βουλευτές οι οποίοι ε, θέτουν τις ίδιες ερωτήσεις διαρκώς, οι οποίες ίδιες ερωτήσεις παραμένουν διαρκώς αναπάντητες. όλα αυτά εγώ θα θέσω πάλι την ίδια ερώτηση, διότι πιστεύω ότι αυτό θα επηρεάσει και τις συζητήσει για τις επόμενες εβδομάδες και τους μήνες. Σήμερα λοιπόν, κυρία Άσκη, μας είπατε και πάλι ότι έχουμε μια καλύτερη προστασία δεδομένων. Από πότε καλύτερη, καλύτερη από το 2001 με τις επιθέσεις ε, ε, που ανέλαβαν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε χωρί να μα ενημερώσουν, μάλλον με την παρέμβαση που ανέλαβαν οι Ηνωμένε Πολιτείε χωρί να μα ενημερώσουν. Από πότε καλύτερα, γιατί τώρα βλέπουμε ότι οι χώρες ακόμη αρνούνται να εξασφαλίσουν αυτή την προστασία των δεδομένων. Μας λέτε δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Ναι, ποια κενά ακριβώ. Γιατί πολλές φορές εδώ ρωτήσαμε να μας δώσετε στοιχεία, αποδείξεις για την ανταλλαγή αυτών προσωπικών δεδομένων, πώς εξασφαλίζεται την προστασία των πολιτών της Ευρώπης. Πώς γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων με προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτικών. Ούτε μία απόδειξη, ούτε ένα στοιχείο δεν μας έχετε δώσει. Δέκα μέρες τώρα, πριν από την υπογραφή στις 30 Δεκεμβρίου της Συμφωνίας, πολλές δηλώσεις δημόσιες και όχι μόνο στην ε, Γερμανία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη φαντάζομαι έλεγαν ότι ε, το SWIFT έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τα λοιπά, αλλά όταν ρωτήσει κανείς τις αρχές που πραγματικά εφαρμόζουν τις υπηρεσίες, που πραγματικά εφαρμόζουν το SWIFT, η απάντηση είναι «Ε, όχι, τελικά δεν μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα». Πείτε μας λοιπόν σε τι έχουμε εμείς κερδίσει. Και πείστε μας ότι δεν διαθέτουμε ε, άσκοπα και ανέμελα τις, ε, τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μας χωρίς καμία σκοπιμότητα, χωρίς καμία, κανένα κέρδος, χωρίς κανένα αντάλλαγμα από τους Αμερικανούς. Επίσης, δεν θέλω να πω ότι το SWIFT, όπως και τα προσωπικά δεδομένα, με ενοχλούν ως προς το θέμα, όχι μόνο δεν έχουμε αντάλλαγμα, αλλά και ως προς ότι δεν έχουμε περισσότερη ασφάλεια, αλλά και ως προς τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να έχουμε ε, προωθήσει και μέσα από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Βλέπω ότι δεν υπάρχει καλή βάση για συνεργασία σε συνθήκες εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πολλές είναι οι επιφυλάξεις και η επιφυλακτικότητα ε, στα όλα θρεμπόριο βάρος των ανθρώπων, των γυναικών, τα εγκλήματα κατά των παιδιών. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία ενδεχομένω, όμως βλέπετε υπάρχει και μια νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως η νέα Προεδρία να μας βοηθήσει να μελετήσουμε διεξοδικά τα θέματα αυτά. Την ε, Πέμπτη έχουμε να συστήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Στον αγώνα για την καταπολέμηση τρομοκρατίας δυστυχώς έχουμε λησμονήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό μαζί με άλλα θα πρέπει να είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά. Ευχαριστώ. Άλλοι δύο συνάδελφοι έχουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι θα πρέπει στις 4 η ώρα να πάει η προσκεκλημένη μας η Νομική Επιτροπή. Οπότε, σύντομη παρακαλώ. Κυρία Υπουργέ, ο κύριος Μπρόντος, δεν ξέρω αν είναι εδώ, ήρθατε έτοιμοι, έτοιμοι να απαντήσετε αυτό το οποίο θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Εγώ τώρα ρώτησα μια εβδομάδα, αλλά δεν πήρα απάντηση, γι' αυτό ρωτώ. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης δεν είναι βάρος στον χάρτη μελετών δικαιωμάτων, από τον οποίο η Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτοξαιρεθεί όπως και άλλες χώρες η αυτοεξαίρεση αυτή θα συνεχίσει να ισχύει τώρα εν ώψη της ε, ε θέσεως τη της συνθήκης Λισαβόνας. Ελπίζω ναι, γιατί νομίζω ότι απειλούνται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στη χώρα μου. Δεύτερον, κάτι μα είπατε για κοινή νομοθεσία και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Αγγλία, Ουαλία και άλλε δύο οντότητε. Ε, κάνουμε στάξει στο στη χώρα μα έχουν άλλο, άλλο σύστημα. Τι θα γίνει. Θεωρείτε ότι θα πρέπει εμείς να χάσουμε ε, αυτή, αυτή τη διαφορετικότητά μας όσον αφορά το, την ένωμη τάξη. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, δύο σημαντικές ε, γραμμές όσον αφορά την υποστήριξη της ε, συμφωνίας ανάμεσα ΕΕ και ΕΕ. Η πρώτη είναι ότι είναι προσωρινή η συμφωνία και η δεύτερη είναι ότι είναι ουσιαστική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και βασίζεται κυρίως σε αυτό που μας είπε και η έκθεση για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ψυχρά αυτά τα δύο συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο νομίζω πως δεν είναι ισχυρό σημείο. Είναι μάλιστα αρκετά αδύναμο και την τελευταία περασμένη εβδομάδα μάθαμε πω τελικά οι εννέα μήνες της προσωρινής συμφωνίας ε, καταλήγουν σε πέντε χρόνια αποθήκευση των ε, στοιχείων μα σε μια βάση δεδομένων που έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένε υποθέσει ε, έρευνα. άρα δηλαδή δεν είναι προσωρινή συμφωνία εννέα μήνων, είναι μια συμφωνία πέντε ετών. Φυσικά τα στοιχεία τα οποία θα, θα συλλεγούν θα θα παραμείνουν αποθηκευμένα για πέντε χρόνια. Άρα λοιπόν με κάποια έκπληξη συζητάμε αυτές τις πληροφορίες και ίσως με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου, αν αυτές οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει σε συμφωνία με τους πυρογνώμονες το συνθήκες της Λισαβόνας, όπως διαρκώς ζητούσαμε από εδώ, θα είχαμε κι εμείς σημειώσει τη δική μας διαφωνία ε, σε σχέση με αυτά τα μειονεκτήματα τη εν λόγω συμφωνίας. Άρα λοιπόν δεν είναι προσωρινή ε, γιατί ο τη ε, ξεπερνά κατά πολύ του εννέα μήνε και θα πρέπει να δούμε τις πρακτικές που θα θεσπιστούν εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε με τις Αμερικανικές Αρχές από αυτές τις βάσεις. Και σε σχέση με το δεύτερο ισχυρό σημείο, λέει πολλές φορές, αναφέρεται μάλλον η έκθεση Γ.Ε.Π. για να πούμε ότι αυτή, η συμφωνία θα, είναι, θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εμείς το συζητήσαμε Ε, συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμη η έκθεση αυτή, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ πιστική από πρακτική άποψη. Εμεί έτσι κι αλλιώ μπορούσαμε να δούμε μόνο το κομμάτι που δεν είναι εμπιστευτικό. Εγώ δεν νομίζω πως υπάρχουν αρκετές ε, εγγύησεις, είναι απλά προφορικές. Στην πράξη δεν υπάρχουν εγγύησεις. Άρα λοιπόν αυτές οι, αυτές οι δύο ισχυρέ υποτίθεται γραμμές της συμφωνίας SWIFT ε, καταραίων. Εμπιστοσύνη λοιπόν χρειάζεται εδώ, μας ζητάτε. Αλλά ακριβώς αυτό εμείς δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας SWIFT. Άρα λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους να εμπιστευτούν μια συμφωνία που δεν τη διαπραγματεύτηκαν οι εκπρόσωποι τους στο Κοινοβούλιο. Και νομίζω πως αυτό είναι πολύ σοβαρό. Υπουργέ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Αλλά ασφαλώς θα αντιληφθείτε ότι έχω ήδη απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και όταν επαναλαμβάνονται χάνω χρόνο ως προς την απάντηση άλλων ερωτήσεων. Για το SWIFT. Λοιπόν. Το, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν πρέπει ναι ή όχι να θέσουμε ένα τέρμα στη χρηματοδότηση εθνούς τρομοκρατίας. Η απάντηση για μένα είναι ναι. Δεν μπορεί κανείς να ε, διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια εφόσον δεν έχει χρήματα στη θέση του. Το σύστημα όμως το χρηματοπιστωτικό επιτρέπει να περνάνε από τη μία στην άλλη οι τρομοκράτες. Όποιος έχει στα χέρια του μία πιστοτική κάρτα ξέρει πώς δουλεύουν, πώς λειτουργεί αυτό το, το σύστημα. Εάν πάρει κάποιος τα στοιχεία της ε, πιστοτικής σας κάρτας και πάει στη Δαμασκό να αγοράσει διαμάντια, το δικό σας όνομα θα φανεί στον κατάλογο της τρομοκρατίας και θα εμπλεκεί σε όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα ενημέρωσης για τα ζητήματα αυτά για τις συναλλαγές αυτές και πρέπει να, αντάλ ε, να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες μας και να αντιδρούμε έτσι ώστε να μην υπάρχει χρηματοδότηση η υποψία χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η προσωρινή συμφωνία ε, έτυχε ιδιαίτερα σοβαρής επιτήρησης, παρακολούθησης ως προς τα στοιχεία που θα μπορούσαν να διαβιβαστούν και ως εκ τούτου ναι, μπορεί κανείς ρητορικό πως να πει δεν ήταν νεάμινη η διάρκειά της αλλά πενταετής ε, αλλά ούτως ή άλλως ήταν ε, όντως εννεάμινη η συμφωνία αλλά νεαμινη η διατήρηση των στοιχείων για πέντε έτη ή το ένα επιχείρημα ή το άλλο. Ε, ό,τι και να πει κανεί ω προ τη διάρκεια, το βασικό είναι ότι προσπαθούμε χάρη στο SWIFT να αποφύγουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να χρηματοδοτούν τους, να χρηματοδοτούν τις τρομοκρατικές ενέργειες με τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Αυτή ήταν μια βάση νομική, ένα σύστημα ε, που βρήκαμε για να έχουμε αυτή τη συνεργασία για την ανταλλαγή δεδομένων με τις ΗΠΑ, που είναι πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του SWIFT. Για ένα πράγμα επέμεινα εγώ, ακριβώς αυτό. Να αγωνιστούμε για την πάταξη της τρομοκρατίας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διάσταση. Για δε τη συμφωνία, βεβαίω θα την υποβάλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξ αρχή ήταν η πρόθεσή μα αυτή. Ε, τρέφω απόλυτο σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αντιληφθείτε κι εσεί ότι μα πιέζει ο χρόνο. Εν τέλει όμω νομίζω ότι επιτύχαμε. Την αποστολή μας ο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ρωτήθηκε εάν θα εφαρμοστεί για, την, ε, για το Ρωμανό Βασίλειο και τι άλλε χώρε που έχουν επιλέξει την αυτοεξαίρεση. Νομίζω ότι μπορεί, χωρίς καμιά δυσκολία, να διαφυλαχθεί για το μέλλον το βρετανικό νομικό σύστημα. Φυσικά κάποια θέματα ε, αρμοδιότητα, κάποια συστήματα αρμοδιότητα δεν μπορούν να μεταφερθούν, να εκχωρηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ε, Μεγάλη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Αντιληπτό και αυτό. Και από την άλλη, πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να ε, κάνουμε ακόμη περισσότερο σεβαστή την ε, σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν κυρώσει τόσα πολλά κράτη-μέλη. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από δικολαβικά επιχειρήματα για να μην εφαρμόζουμε, για να μην προστατεύουμε αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες Ξέρω ότι είναι περιπλοκή κατάσταση, αλλά απαραίτητο για μένα είναι και στο πίσω τη ευρωπαϊκή μα συνεργασία να γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίε. Ελπίζω να έχω απαντήσει όλε σα τι ερωτήσει, χωρί να είμαι βέβαιο ότι ικανοποίησα του πάντε, αλλά δεν ήρθα για να σα χαϊδέψω τα αυτιά. Η πρόεδρο. Λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο γιατί έχουν στήσει το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Κυρία Σκ, σα ευχαριστώ για την διαθέσιμότητα να έρθετε να μας μιλήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι θα πρέπει να αποχωρήσετε. Σας ευχαριστώ και πάλι στα αγγλικά, κυρία Σκα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και αν μου επιτρέπετε, καλά Χριστούγεννα. Ήταν σκληρή δουλειά όλο αυτό τον σκοτεινό Νοέμβριο και θα είναι και το Δεκέμβριο. Ελπίζω να συνεχίσετε τις καλές σας συζητήσεις εγώ στηρίζομαι στην στήριξη του Κοινοβουλίου και για την Άνοιξη. colleagues, now we Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Προεδρία, Σουηδική Προεδρία και αποτελέσματα της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Μεταξύ μας βρίσκεται ο κύριος Τοπίας Μπίλστρομ, Υπουργός για τη μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου της Σουηδίας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπίλστρομ, που ήρθατε που στη διάθεσή μας για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις μας. Θα ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή όχι τι έχετε να μας πείτε για τη δουλειά των τελευταίων μηνών και περιμένουμε τα αποτελέσματα στον τομέα της μετανάστευσης, τις εξελίξεις μάλλον στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Πριν από λίγε εβδομάδε στο Στρασβούργο, κύριε Πρόεδρε, τότε που συζητήσαμε το πρόγραμμα τη ε, Στοχόλμη, επικοινωνήσαμε, αλλά με μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε και σήμερα. Ε, θα πρέπει επομένω να κάτσουμε και να δούμε τι έγινε κατά την Σουηδική Προεδρία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το φθινόπωρο ήταν φορτωμένο από πάρα πολύ ενδιαφέροντα ε, γεγονότα. Είχαμε σημαντικέ θεσμικέ εξελίξει όπω την θέση και τη Λισαβόνα. Τώρα επομένω μπορούμε να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας και τον ενδιαφέρον μας στο, στο, στο, στο τι θα κάνουμε πέρα πέρα. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρο, ο πρόεδρος, δεν είναι εδώ, αλλά θα πρέπει να συνηθούμε για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια επί τη βάση του προγράμματος της ε, Στοκόλμης. Η Συνδίκη της Λισαβόνας πάντως επιφέρει τις πολύ σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια, ιδίω όσον αφορά το πόσο έχει αναβαθμιστεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ διαφορέ στην συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Όμω, ήδη είχαμε κάποιε θετικέ εμπειρίε σχετικά με αυτό κατά την ε, Προεδρία μα. Εγώ τώρα θέλω να σα πω για κάποιε επιτυχίε που σημειώσαμε όσον αφορά το άσυλο αλλά και τη μετανάστευση κατά την Προεδρία μα. Πρώτα-πρώτα κάτι το οποίο ήταν υψηλή προτεραιότητα της Προεδρίας μας και μιλώ για την ε, πρόσβαση χωρίς θεός διαβατηρίου ε, από τρεις χώρες προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σερβία, Μαυροβόνια και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουμε βιομετρικά διαβατήρια και αυτό από τι 19-12 του 2009 θα τεθεί σε ισχύ απόφαση. Να, ένα ωραίο χριστιανικό δώρο που θα μπορούσε κανεί να πει προ του ε, λαού εκείνου, οι οποίοι τώρα θα μπορέσουν να γιορτάσουν ε, τα Χριστούγεννα με του συγγενεί και φίλου που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά τα πλαίσια να μην ξεχνούμε άλλα δύο χώρε ε, οι οποίε έχουν κάνει σημαντικά βήματα προ την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε αυτό το, το κοινό ανακοινωθέν Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θέλουμε να αφαιρούμε την Αλβανία και Βοσνία Τζεκοβίνη για να προβούν εις, ε, τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Για να μπορούν και αυτές οι χώρες να έχουν πρόσβαση χωρίς διαβατήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω τώρα δύο λόγια για τη Λισαβόνα, ακριβώς ε, όπως θα διαμορφωθεί μια πορεία για την επόμενη πέντα αιτία. Ξεκινώ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα σχετικά με αυτά και πριν από λίγε εβδομάδε ε, κάναμε μια συζήτηση πάρα πολύ μεστή στο, στο, στο Στασβούργο. Είχαμε ε, 30 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου το Συμβούλιο των Υποθέσεων και σημειώθηκε μια ε, σύμφωνη γνώμη των, των ε, κρατών μελών και πάμε για έγκριση στο, στη συνάντηση 10-12 Δεκεμβρίου. Είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Τώρα μπορούμε να έχουμε μια πολιτική για άσυλο μετανάστευση και ξεκινάμε λέγοντα ότι είναι δυνατόν όλοι οι εμπλεκόμενοι να ε, έχουν καλύτερο πλαίσιο στο οποίο να κινηθούν για, την μετανάστευση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούμε να καλύψουμε τι ανάγκε των κρατών μελών, να μπορέσουμε να είμαστε επίση και συμμορφούμενοι με την της Σαββόνας. Τώρα, η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σε αυτό το πρόγραμμα. Τα δε τα μέτρα όπως εταιρική σχέση, όπως κινητικότητα, όλα αυτά θα έχουν στρατηγική σημασία και θα πρέπει επομένως να λάβουμε υπόψη αυτές τις συνεργασίες και τις θετικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης επίσης θα φροντίσει για το να υπάρξει μια πολιτική ανάσχεση της λάθρο μετανάστευσης. Πάρα πολύ σημαντική η δουλειά, πάρα πολύ σημαντική και η Frontex ε, σε αυτήν την, ε, την υπόθεση, σε αυτή την πορεία. Θέλουμε μια ισορροπία, θέλουμε κάποια μέτρα ασφάλειας τα οποία να, να, αλλά χωρίς να παραβλάψουμε, να βαρύνουμε, να ενοχλήσουμε τους νόμιμους μετανάστες. Άρα θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε και τους ε, αφεντικούς ελούντες άσυλο, να μην ε, θίξουμε το, το πλαίσιο που βοηθά ε, τους ανήλικους που ζητούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται αλληλέγγυα στάση μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών μελών και μεταξύ ε, των τρίτων χωρών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι θέλουμε να βρούμε κάποιες ε, λύσεις βιώσιμες, κάποιες λύσεις διαρκής σε σχέση με ε, το αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο της μετανάστευσης. Τα κράτη-μέλη έχουν φυσικά ζωή πολλών μεταναστών. Χρειάζονται επομένω μία βοήθεια. Ε, να έχουμε κάποιο capacity building, δηλαδή να έχουμε τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Στην κέντρη της Λισαβόνας επίσης μόλις τεθεί σε ισχύ θα μας δώσει πολλά εργαλεία. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης πάντως επιβεβαιώνει το ότι είχαμε ε, μέχρι το 2012 τάξει κάποιους στόχους. Αυτοί συνεχίζουν και ισχύουν. Και έτσι επίσης επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια κοινή ράχο κοκαλιά ε, στο τι σε κάθε κράτο μέλος και ότι ο καθένας αυτούς που ετούνται άσυλο θα τύχουν ευμένους υποδοχή, θα τύχουν εξέταση ε, ε, η οποία θα είναι ομοιογενή σε όλα τα κράτη-μέλη, όπου και αυτοί να επιβάλλουν την αίτηση. Όλα αυτά τα τονίζουμε και τονίζουμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε την εξωτερική διάσταση. Υπάρχει μια πάρα πολύ στενή σχέση μεταξύ εξωτερικών σχέσεων και της δουλειάς που γίνεται στο εσωτερικό για ασφάλεια δικαιοσύνη και ελευθερία. Όλα αυτά ε, υπάρχουν στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο. Και τέλος εβδομάδας θα εγκριθεί ελπίζουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα το οποίο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα το εγκρίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα μπορεί να προσφέρει πρόγραμμα δράση για την υλοποίηση του προγράμματο τη Στοχόλμη. Μάλλον αυτό θα γίνει αρχά του επόμενου έτου. Κύριοι βουλευτέ, όπω είπαμε πριν από μερικού μήνε, επιβεβαιώσαμε το πρόγραμμα τη Στοχόλμη για το ότι Μέχρι το 2012 θα έχουμε ένα κοινό σύστημα για άσυλο και μετανάστευση, πάρα πολύ φιλόδοξο βέβαια αυτό ο στόχο. Και εμεί πάντω κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν ούτω ώστε τα πράγματα να πάρουν αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό σα λέω ότι με μεγάλη μα χαρά τώρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων. Ε, υπάρχει κάποια υπηρεσία υποστήριξη και θεωρούμε ότι σε συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα θα συγκροτήσουμε αυτή την υπηρεσία, ούτως ώστε να υπάρχει μια αντίστοιχη νομοθεσία πλαίσιο που να μας βοηθήσει με αποτελεσματικό τρόπο και έτσι να υπάρξει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι αυτές εξελίξεις θετικές και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε συνεργασία αποδοτική μεταξύ ε, των μελών. Αυτό πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου. Τώρα, αυτή η υπηρεσία στήριξης θα εδρεύει στην Βαλέτα και δουλεύουμε ούτω ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης πανκοινωτικό, πανενωσιακό και να υποστηρίζεται από το ταμείο ε, το οποίο προβλέπεται να, που έχει δημιουργηθεί για την μετανάστευση. Ελπίζω να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που ελπίζουμε να αρχίσει να τρέχει όσο γίνεται νωρίτερα του χρόνου αυτό, αυτή, αυτή η υπόθεση, αυτή η πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τι άλλε προτάσει για τροποποίηση κάποιων νομοθεσιών που αφορούν το κοινό σύστημα ασύλου, είναι πρώτη ολόκληρη δέσμη μέτρων. Ε, έχουμε σημειώσει και εδώ σημαντική πρόοδο και κάποιες προτάσεις είναι αρκετά περίπλοκες, πολλές φορές εξαρτώνται από κάποιες άλλες πολιτικές αποφάσεις. Νομίζω ότι το έργο μας θα είναι ευκολότερο, πάντως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει όλες τις προτάσεις που αφορούν την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του κοινού συστήματος ασύλου. Και έτσι Μπορούμε τώρα να δούμε οι ελιοσχετιζόμενες αυτές προτάσεις πώς μπορούν να προωθηθούν όλες μαζί. Τον Ιούνιο είχαμε κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο για την Μεσόγειο. Είχαμε την λήψη κάποιων μέτρων. Άρα τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μέτρα δυναμικά, κατά το οποίο τον Οκτώβριο το ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα τρία δεσμικά όργανα συμφώνησαν να υπάρχει αυτό το γραφείο υποστήριξη σε συνέχεια και η υλοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Είπαμε ότι αυτό θα εδρεύει στην Μάλτα και θα μπλακούν μια σειρά κράτη-μέλη. Έχουμε αρχίσει διάλογο και συνεργασία με χώρες προέλευσης, με χώρες διέλευσης. Εξού και η συνεργασία με την Τουρκία πριν από ένα μήνα. Και έτσι θέλουμε να υπάρξει διάλογος για θέματα της μετανάστευσης και με την Τουρκία και να αρχίσουν να ξαναρχίσουν οι διακοπές διαμοτεύσεις για κάποιο είδους αποστολή μας εκεί. Θέλουμε να βρεθεί βιώσιμη λύση. όλοι αυτοί οι οποίοι διακινούν τη ζωή του για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο. Οπότε με το πρόβλημα τη ε, Στοκόλμη τώρα έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε το μέλλον. Για άλλη μια φορά σα ευχαριστώ πάντω. Σα ευχαριστώ για την τόσο θετική συνεργασία. Χωρί τη θετική αντιμετώπιση που είχαμε από εσά, δεν θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε την υπηρεσία αυτή ε, της, της, της δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα που είναι τόσο φιλόδοξο όσο ο τη Στοκχόλμη. Περιμένω πώ και πώ τώρα τι τυχόν ερωτήσει που έχετε. Σα ευχαριστούμε κυρία Μπίλστρομ. Συναρπαστική και σημαντική η περίοδος που διανύσατε, κυρίως σε σχέση με την ε, θεωρήσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εγώ θα πρότεινα να έχουμε δύο-τρεις γύρους ερωτήσεων και, μάλλον, ερωτήσεων και μετά απάντηση της δικής σας, γιατί έχουμε αρκετούς συναδέλφους που θέλουν να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Και πρώτα ο κύριος Μπουζουτήλ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας ε, τον θαυμασμό ε, μου, γιατί πήγατε την κόρη σας ε, στο Συμβούλιο των Υπουργών την περασμένη εβδομάδα. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα ποιοτικού χρόνου με την οικογένεια. Αν και δεν νομίζω ότι εγώ θα είχα στο μυαλό μου ένα συμβούλιο του, ένα, μια συνεδρία του Συμβουλίου ως ποιοτικό χρόνο για να περάσουμε τα παιδιά μου. Εν πάση περιπτώσει να σας συγχαρώ για τα όσα καταφέρατε που καταλήξατε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ασύλου. Ήταν σημαντικό επίτευγμα και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό. Αλλά επίσης ξέρετε κύριε Υπουργέ πως το πακέτο περί ασύλου αποτελείται από διάφορες άλλες νομοθετικές προτάσεις και η Προεδρία ίσως βολικά ακολούθησε μάλλον φέρεσε το πιο εύκολο θέμα από το πακέτο, όπου σωστά όπως φάνηκε πίστεψε πως θα πετύχει συμφωνία. Ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι τι γίνεται με τις υπόλοιπες νομοθετικές προτάσεις του πακέτου περί Πώς βλέπετε να συνεχίζεται η υπόθεση αυτή τα επόμενα χρόνια, γιατί η εντύπωσή μου είναι πως το πακέτο αυτό είναι πλέον είναι πολύ μεγάλο, πολύ περίπλοκο ε, για να επιτευχθεί συμφωνία τώρα κοντά. Να στραφώ και σε δύο άλλα ε, σημεία. Αναφέρεται το θέμα της αλληλεγγύης και επίσης αναφέρετε την εκκίνηση ενός πιλωτικού προγράμματος για την εσωτερική επανεγκατάσταση ε, χωριστά. Επίσης αναφέρατε και την εξωτερική επανεγκατάσταση, δηλαδή το, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εξωτερική Επανεγκατάσταση. Για την εσωτερική επανεγκατάσταση και το σχετικό πρόγραμμα έχω την εντύπωση ότι 6-7 κράτη-μέλη από τα 27 έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρείτε πως αρκεί και τέλος, για το θέμα της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Αναφέρατε ότι έχετε πολύ, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρα επίσκεψη στην Τουρκία. Ε, από ό,τι κατάλαβα, Υπουργέ, χρειάστηκε να επισκεφθείτε και τη Λιβύη. Ποιο ήταν τα αποτελέσματα της απόπειρας να πάτε στην Λιβύη και πώς βλέπετε τη συνεργασία με τη χώρα αυτή για το θέμα της μετανάστευσης. Ευχαριστούμε κυρία Γκόντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ε, Σουηδική Προεδρία. Ήταν όντως πολύ έντονη περίοδος και θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Να αναφέρω ότι υπάρχει ε, καθεστώς ε, χωρίς θεωρήσεις για τις ε, τρεις ε, χώρες, ε, το Σερβία κτλ. Και ελπίζουμε πως σύντομα θα έχουμε το ίδιο καθεστώς και για την Αλβανία και την Βοσνία Ριζεγοβίνη όπως είπατε και εσείς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της αλληλεγγύης. Είδαμε στην συμφωνία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των ευρωπαϊκών θεσμών και τις απόψεις των κατών μελών. Εγώ θέλω να ρωτήσω μάλλον να ακούσω περισσότερα σε σχέση με τις εμπειρίες τους. Πώς περιμένετε να γεφυρωθεί αυτό το κενό. Πώς μπορούν ε, δηλαδή να προσεγγίσουν ε, οι απόψεις σε σύμφωνα με τις πρόσφατες προσπάθειες που κάνατε όσον αφορά την επανεγκατάσταση, γιατί νομίζω πως θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Το άλλο που αναφέρατε δηλαδή η, διαδικασία, η ενιαία διαδικασία ασύλου. Ε, υπάρχει διαφορά σε σχέση με την προσέγγιση των αρχών μας. Αρκετά μεγάλη όταν δούμε την πρακτική κάθε χώρας. Πώς βλέπετε το μέλλον αυτές τις διαδικασίες και ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον. Τρίτη ερώτηση. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναζητούν διεθνή προστασία. Οι πιθανότητες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι να περάσουν παράνομα τα σύνορα τις περισσότερες φορές. Πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ζητήσουν άσυλο πριν να θεωρηθούν παράνομοι μετανάστες είναι ένα θέμα για το οποίο νομίζω θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η κυρία σα σας ευχαριστώ. Νομίζω πω για το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη έχουν γίνει κάποια πολύ καλά βήματα από τότε που έκανε την ανακοίνωσή τη, η Κομισιόν κινήθηκε προς καλή, κινηθήκαμε προ καλή ε, κατεύθυνση και επίση υπάρχουν ε, εξελίξει ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί. Έχω όμω και κάποιε επικρίσει, ε, δεν είναι όλα τέλεια στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη, όπω τα ήθελα εγώ. Για παράδειγμα για το Frontex και τα συμφωνίε επανεισδοχής οι διαπραγματεύσει που γίνονται με την Τουρκία και τη Λιβύη, για παράδειγμα, εγώ βλέπω να λείπει η διαφάνεια. Πρέπει να ρωτήσουμε κάθε φορά τι συζητάτε με τη Λιβύη, ας πούμε. Θα έχουμε το, ε, να έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε τι συμβαίνει εκεί και να γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνει το Frontex στις επιχειρήσεις του. Και αυτό Αυτά για την ώρα δεν υπάρχουν. Θα θέλαμε να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη διαφάνεια. Και ούτε αναφέρεται στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη μέχρι στιγμή. Ίσως αυτό θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξει. Στους ίδιους τομεί όπου μιλάμε για συνεργασία με τρίτες χώρες, μάλλον το Συμβούλιο και η Σουηδική Προεδρία τη Λάγια συνεργασία με τρίτες χώρες, αφορά αυτό μόνο αποτελεσματική επιστροφή των παράνομων μεταναστών, αλλά δεν γίνεται πουθενά λόγος, για παράδειγμα, για προδιαγραφές ε, ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων, ε, σεβασμό αυτών κτλ. Δηλαδή, δεν είναι το πάνη αποτελεσματικότητα. Θέλουμε, ναι, εντάξει, να τους επιστρέψουμε τους μετανάστες, αλλά να υπάρχουν και κάποια στάνταρ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες όπου επιστρέφουν. Θα πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσέχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ίσως να μπορούσαμε και να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες να φτιάξουν ε, περισσότερο την κατάσταση. Δύο ακόμα παρατηρήσει. Το πρόγραμμα στο Στοκχόλμη λέτε για κοινή προσέγγιση προ τρίτε χώρε που δεν συνεργάζονται μέσα στο πλαίσιο τη επανεισδοχή. Τι σημαίνει ακριβώ αυτό, Δηλαδή, ποια θα ήταν μια κοινή προσέγγιση. Α πούμε όταν μιλάμε για την Τουρκία, δεν υπάρχουν, θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξή τη αν δεν υπάρχει πλέον επανεσδοχή. Ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κοινή προσέγγιση. Και μετά λέτε ότι το Frontex θα πρέπει να έχει περισσότερη επιχειρησιακή συνεργασία με τρίτες χώρε. Φαντάζομαι πω γνωρίζετε την απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του και που έλεγε ότι το Frontex δεν θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τρίτε χώρε ή να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις από μόνο του. Δηλαδή, τι ακριβώς ε, εννοείται όταν μιλάτε για επιχειρησιακή συνεργασία. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις πριν να περάσουμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας θα απαντήσω στον κύριο Μπουζούτσιλ. Τον ευχαριστώ για τα ευγενικά του λόγια για την παρουσία της χώρα μου στη συνεδρία του Συμβουλίου. Δεν φανταζόμουν ότι θα προσελκούσε τόσο πολύ το ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Εν πάση περιπτώσει, καλή οργά παρά ποτέ. Πρέπει το παιδί κάποια στιγμή να ε, έρθει αντιμέτωπο με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Καλή οργά παρά ποτέ λοιπόν. Τώρα για το άσυλο και το Συμβούλιο, το, το, τα θέματα του ασύλου και τη εργασία του Συμβούλιο. Εμείς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τις διαδικασίε. Όπως γνωρίζετε όμω κύριε Μπουζούτιλ και οι λοιποί συνάδελφοι, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσει απόψε μεταξύ των κρατών μελών, όπως και μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή. εν προκειμένου ότι ήδη το γραφείο ε, συντονισμού για το άσυλο μπορεί να αποτελέσει μια πολύ χρήσιμη λύση γιατί θα επιτρέψει την ουσιαστική συνεργασία στα θέματα του ασύλου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόοδος που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής πιστεύω. Για δε το άλλο ζήτημα που θέσατε, πόσες χώρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πιλωτικό πρόγραμμα που, λαμβάνει χώρα, που θα λάβει η χώρα μάλλον στη Μάλτα. Φυσικά τίθεται το, το ζήτημα σε ποιο βαθμό έχει... Ε, μάλλον από ποιο όριο κρίνεται επαρκή η συμμετοχή σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Για μένα ουσιαστικό κριτήριο είναι το ότι λαμβάνει η χώρα ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα. Και μετά υπάρχουν τα εσωτερικά κριτήρια της κατανομής των ατόμων που ε, χρήζουν προστασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω τα τελικά πορίσματα αυτού του πιλωτικού προγράμματος. Για δε τη Λιβύη, τόσο εγώ όσο και ο Αντιπρόεδρος ε, Μπαρό επισκεφθήκαμε τη Λιβύη πέρυσι για να συναντηθούμε με την κυβέρνηση. Εκεί στο πλαίσιο των, ε, της συνεργασίας μας με τη Λιβύη. Όμως ε, έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση η απάντηση της κυβέρνησης και τελικά δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ για να συναντήσουμε τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος μάλιστα έτυχε να είναι και άρρωστος. Για την κυρία Τζόνς. Συμμερίζομαι τις απόψεις, είναι πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις σας. Μιλήσατε για την Αλβανία και τη Βοσνία ριζεγοβινη Το όντι είναι κράτη αυτά τα οποία θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή της, ε, ε, του καθεστώτους της θεώρησης διαβατηρίων, ώστε να είναι έτοιμα όταν έρθει η ώρα. Εμείς, έχοντας τα σπίση στο σύστημα για τις εξαιρέσεις, περιμένουμε να δούμε τώρα τις θέσεις του Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή και θέλουμε μια στρατηγική επιτροπή, μια επιτροπή η οποία θα μας δώσει αποτελέσματα για το σύστημα αυτό. Από τη θέσπιση της και μετά μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Τα προβλήματα σε σχέση με το άσυλο βέβαια είναι πολλά. Τις ε, λεπτές έννοιες διακυβεύονται και επισημαίνω ότι υπάρχει στο κεφάλαιο το άσυλο μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, το οποίο διαβάζει το οποίο μιλάει για τα εξωτερικά σύνορα και αναφέρω στα αγγλικά, σας διαβάζω, ότι το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να ε, αποβαίνει εις βάρος ανθρώπων που έχουν ανάγκη ε, και είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Εκεί θα πρέπει να προστατευθούν ε, τα δικαιώματά τους όπως και τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές το κείμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτική δήλωση, μια διακήρυξη απόλυτα σαφή. Λέμε με απόλυτη σαφήνεια ότι πρόκειται για θέματα στα οποία πρέπει να ε, δουλέψουμε σκληρά. για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και θέλω να ευχαριστώ την κυρία Βουλευτή για τι παρατηρήσει τη. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε, χωρί να συμφωνούμε βέβαια πάντοτε. Οι παρατηρήσει ε, και για το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη ε, είναι πάντοτε πολύ χρήσιμε. Και είναι απαραίτητο να ε, διαχειριστούμε τι μεταναστευτικέ ροέ, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα. Για δε τις συμφωνίες και της, ε, τη συνεννόηση με τα γειτονικά μας κράτη. Έχουμε πιστεύω την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Είχαμε συζητήσεις, ή μάλλον μη συζητήσεις με τη Λιβύη, γιατί στην Τουρκία είχαμε σημαντικές συζητήσεις με την ε, τουρκική κυβέρνηση. με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ατόμων ε, των προστασία μέσα στην Τουρκία την ίδια. Και, δε, και επίσης μέσα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα αυτή την πτυχή. Στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε αυτά πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και πρέπει σε κάθε μας ε, συζήτηση να τα θέτουμε ως κριτήριο. Για την κοινή προσέγγιση, η Frontex έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό επίσης πιστεύω. Εάν θέλουμε να ε, καταλήξουμε σε μια καλή αποτελεσματική δουλειά, σε ένα καλό αποτέλεσμα, πρέπει να βελτιώσουμε την Frontex χρειάζεται περισσότερη δουλειά και όχι λιγότερη, περισσότερο συντονισμό και όχι λιγότερο για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Η Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Έξι συναδελφοί έχουν στήσει εδώ μεταξύ το λόγο. Έχουμε ακόμη δύο γύρου συζητήσεων. κυρία Βίλστρομ, Ταβάρε και Αλβάνο. Φίξτρομ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα εδώ που ήρθατε σε αυτή την Επιτροπή και έχετε έρθει πολλές φορές. Είχαμε σημαντικές συζητήσεις μαζί σας. Ως μέλος του Κοινοβουλίου πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με τους ειδικοί Προεδρία και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σκληρή δουλειά που κάνατε. Ήρθατε πολύ συχνά ε, να συνομιλήσετε μαζί μας και όλοι σας οι συνάδελφοι έπραξαν το ίδιο. Έχουμε μιλήσει για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις σχετικά και νομίζω πως ε, οι πολίτες ασχολούνται ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά. Πολύ θετική ήταν η ανταπόκριση εν γέννη και πολλές καλές ιδέες έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Και μέχρι στιγμής θελήσατε να ενισχύσετε τα ε, δικαιώματα και γι' αυτό και πιστεύω πως το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα δείξει το δρόμο για να τοποθετηθούν ε, οι ανθρωπιστικές ανησυχίες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Υπάρχουν ωστόσο πολλά προβλήματα που πρέπει ακόμα να επιληθούν. Πρέπει ιδιαίτερα να δουλέψουμε ε, με όσους ε, διακινδυνεύουν την υγεία τους για να μπουν και τη ζωή τους πολλές φορές για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα. Να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους ώστε να είμαστε βέβαιοι πως θα μπορούν να έρχονται εδώ νόμιμα. και να δείξουμε μηνύματα θετικά, καλής βούλησης. Το αναφέρατε και εσείς κύριε Μπίλστρομ. Αυτό είναι ένα βήμα, είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε δυνατότητες για αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορούν δηλαδή να πάνε στην πρεσβεία τους, στην πρεσβεία των κρατών μελών μας ολόκληρο τον κόσμο και να βρουν ένα νόμιμο τρόπο να ζητήσουν άσυλο και να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Τώρα, τον Πίας, εσύ θα ήσουν ε, έτοιμος να Κάνει αυτό που πρότεινε η Άμνεστη, η Διεθνής Αμνηστία, να ζητήσουμε δηλαδή από τους πολίτες να ανοίξουν τις πρεσβείες τους. Να έχει ο κόσμος τα νομικά ε, ε, ε, μέσα στη διαθεσία του που χρειάζεται για να μπορέσει να ζητήσει άσυλο από την Ευρώπη. Αυτός θα ήταν ένας τρόπος για να προσπαθήσουμε να βασιστούμε στην καλή βούληση που ξεκίνησε με την, ε, με την Συμφωνία της Στοκόλμη. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και εμείς ε, θέλουμε να συνεχίσουμε και να υποστηρίζουμε τα όσα εσείς ξεκινήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θα σας, προσπαθήσω να είστε, θα σας προσπαθήσω να σας ζητήσω να είστε σύντομοι, γιατί διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα με το χρόνο μας πάλι. Ο κύριος Σταβάρης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι πολύ επικριτικός για ορισμένε πτυχέ των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη μετανάστευση και πιστεύω πως θα έπρεπε να κινηθούμε προς μια δίκαιη, ρεαλιστική και κυρίως δίκαιη μάλλον και ρεαλιστική πολιτική σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επιμείνουμε στην, ε, στο άνοιγμα και τη διατήρηση νομίμων διόδων μετανάστευσης. Και Γι' αυτό και χάρηκα που άκουσα τον Υπουργό να μιλά, τουλάχιστον εν μέρη, ε, με βάση αυτές τις γραμμές. Η Σουηδική Προεδρία θα πρέπει να επενεθεί για τη δουλειά που έκανε. Και το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Άσυλο είναι ένα σημαντικό βήμα και εγώ θέλω να θέσω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για την επανεγκατάσταση που επίσης έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου. Η επανεγκατάσταση είναι μια μόνιμη λύση, για, ειδικά για πρόσφυγες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Δεν μιλάμε για κάτι το αδύνατο, κάποιο άλλο το πρόβλημα η UNHCR μιλά για 200.000 ε, πρόσφυγες που θα πρέπει να εγκαταστήσονται ετησίως. Οι ΙΠΑ δέχονται περίπου 60.000, άλλες χώρες επίσης ε, δέχονται το δικό τους μερίδιο όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία και ορισμένοι ξεκινούν τώρα όπως η Βραζιλία ας πούμε. Στην Ευρώπη έχουμε μακρά παράδοση. Και ο, και ο για το θέμα αυτό συμφωνεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι ε, για να επιμείνουμε για ένα καλό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για κατάσταση στο κόσμο όμω εκείνος ο οποίος έχει διακινδυνεύσει τη ζωή του στη χώρα του, να μην χρειάζεται να ξαναδιακινδυνεύσει τη ζωή του, προσπαθώντα να διασχίσει τη Μεσόγειο, για παράδειγμα, με σχεδίες. Αλλά αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι ακόμα πρόγραμμα είναι κάποια βήματα μόνο. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μια γραμμή του προπολογισμού που βασικά βοηθά τη χρηματοδότηση των χωρών που υπόσχονται ότι θα δεχτούν και θα εγκαταστήσουν ε, πρόσφυγες. και νομίζω πως αφού έχω συζητήσει εντός του Κοινοβουλίου και με τους συναδέλφους και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα προσπαθούμε να δούμε ποιο θα ήταν το θέμα έτσι ώστε οι νέες χώρες να ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα της εγκατάστασης προσφύγων δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι οι ανθρώπινοι πόροι, είναι η πυρογνωμοσύνη, η οικονομία κλίμακας. Και... Αυτό που θέλω εγώ να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται. Με, τι, πιστεύετε για μια μόνιμη μονάδα που θα εργάζεται για την εγκατάσταση προσφύγων μέσα ας πούμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης Ασύλου ώστε ενδεχομένως να μπορούσαν να εκδίδονται σε προειδοποιήσεις όταν υπάρχουν ανθρωπιστικές κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σύστημα που έχουμε τώρα νομίζω πως δεν ανταποκρίνεται στις επίγουσες αυτές καταστάσεις. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για την κατάσταση προσφύγων που ε, επίσης ε, αφορά το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στήριξης Ασύλου. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Μπίλστρομ κάτι το οποίο ήδη είχα ρωτήσει το Σεπτέμβριο όταν ήρθε ο Υπουργό σα στην Επιτροπή μα. Όμω τότε δεν έλαβα απάντηση. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν τώρα να ακούσω την απάντησή σας. Πριν από λίγο μιλήσατε για ισότιμη μεταχείριση των των άσυλο, το οποίο φυσικά δεν μπορεί παρά να με καθησυχάσει. Όμως αν θυμάστε, φέτος το καλοκαίρι ορισμένε χώρες μέλη έκαναν ε, επαναπατρισμούς τελείως ανώμαλους και δεν επιτράπηκε σε εκείνους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στις ε, βάρκες ε, να ζητήσουν άσυλο δεν, δεν αναγνωρίστηκαν καν, απλώς ε, διώχτηκαν. Είχα κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν και δεν μου δόθηκε απάντηση. Ίσως το Συμβούλιο να μην μπόρεσε να μας πει εμάς τίποτα. Αλλά δεν ξέρω αν ε, στη συνέχεια υιοθετήθηκαν κάποιες προβλέψεις. Ε, εγώ θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι πιστεύετε εσείς. Και πριν από λίγο υπογραμμίσατε την ανάγκη να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση. Μα θα γίνει κάποια αναφορά σε σχέση με θα γίνεται μάλλον διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς που φεύγουν και από μια κατάσταση ε, επίγουσα. Δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ξεφεύγουν από τον πόλεμο ή από διώξεις ε, και σε εκείνη την περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι πάλι μεταχειρι... τους μεταχειριζόμαστε σαν να είναι ε, παράνομοι μετανάστες και διώκονται. Τελευταία ερώτηση, που δεν είναι όμως λιγότερο σημαντική. Άλλοι συνάδελφοι σας ρώτησαν για τη Λιβύη και τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Εσείς είπατε πως δυστυχώς δεν υπήρξαν αρκετές ε, ευκαιρίες για να εμβαθύνεται στα θέματα με τη Λιβύη. Όμως, πριν από τρει εβδομάδες περίπου, ορισμένοι υπάλληλοι τη ε, Σουηδική Προεδρίας είπαν άλλα πράγματα. Είπαν ότι υπάρχουν, ε, ότι έγιναν μάλλον τεχνικής φύση επαφές και ότι αυτές οι τεχνικές φύση επαφές θα εξυπηρετούσαν την εξομάλυση των σχέσεων με αυτή τη χώρα, τη Λιβύη. Και εγώ ρώτησα ξεκάθαρα, μα τι σκοπεύετε Πώς μάλλον σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτές τις επαφές με την Λιβύη. Θα λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η Λιβύη, για παράδειγμα, δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση της Γενέβης. Θα λάβετε υπόψη ε, το γεγονός ότι η Λιβύη, για παράδειγμα, δεν επιτρέπει μέχρι στιγμή σε κάποιους παρατηρητές ε, του ΟΗΕ και να συζητήσει με τους πρόσφυγες και με τους φυλακισμένους. Σας ζητώ λοιπόν να μου απαντήσετε, γιατί για μένα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου μόνο ένα λεπτό. Tack så mycket för ordförande. Än en gång jag skulle bara konferera här ett ögonblick. Jo, först och främst Wikström då. Θα ήθελα να πω, κύριε Μάλκτρομ, ότι όντω είναι πολύ σημαντικό το θέμα της μετανάστευσης για τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης, γιατί μιλάει στον πολίτη Μιλάει στον πολίτη που βρίσκεται έξω από την Ένωση. Για δε τη λάθρο μετανάστευση πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, όπως έλεγα και νωρίτερα, ισορροπία αφενός μεν ελέγχου, αποτελεσματικού ελέγχου στα σύνορα, αφετέρου δε ελέγχου, ο οποίος ταυτόχρονα κάνει σεβαστά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ετών του άσυλου. Στην απάντηση που έδωσα νωρίτερα στην κυρία Γκρόνς και την κυρία Κέλλερ, αναφέρθηκα στα προβλήματα πρόσβασης στο σύστημα. Δεν είναι απλό το πρόβλημα. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να βρούμε μια πιο αποτελεσματική ρύθμιση και ταυτόχρονα απαντώντα τον κύριο Ταβάρης θα έλεγα ότι είναι ίσως πιο εύκολο για μας να, συνεχίσουμε την ε, ε, παράδοσή μας γιατί η Σουηδία έχει ανέκαθεν συνεργασία με τα κράτη προελεύσεως και βλέπουμε ότι όντως ε, φέρνει αποτελέσματα. Γι' αυτό θα θέλαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη ε, προελεύσεως. Για δε ένα ευρωπαϊκό σύστημα συνεργασίας, διερωτώ με θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη και να συμβάλλουν σε αυτό. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν ποσοστώσεις υποδοχής Όταν έχουμε 100.000 άτομα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 100.000 άτομα, το επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να διαχειριστεί κανείς κατά τρόπο αυτόματο. Πρέπει να, προσ... εξασφαλίσουμε την προστασία για τους πιο ευάλωτους, για τους ασθενέστερους, να, τους... να επιτρέψουμε εκείνους που κινδυνεύουν στις χώρες τους ε, και να του προσφέρουμε το άσυλο και την προστασία. Και εδώ απαλώ στον κύριο, κύριο, Τάβαρες. Εμείς με βάση αυτές τις αρχές εργαζόμαστε. Κύριε Τάβαρες, χωρίς να θέλω να υψέλθω λεπτομέρειες, για το γραφείο αυτό γιατί τις λεπτομέρειες θα τις δούμε κατά τη συνεργασία, κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου υπό την ε, Ισπανική Προεδρία. Χωρίς λοιπόν να φέρω νύψη αυτές τις λεπτομέρειες, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε την ανάγκη για συνεργασία όχι μόνο μεταξύ κρατών της Ένωσης, αλλά και κρατών της Ένωσης, ε, μάλλον της Ένωσης αφενός και άλλων κρατών όπως Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά. Όσο πιο πολύ αναπτύσσεται αυτή η διεθνή συνεργασία, τόσο ευρύτερη θα είναι και η προστασία που θα μπορούμε να προσφέρουμε στα πραγματι χρήζοντα άτομα. Και στο ρόλο που θα διαδραματίσουν τα, θεσμικά όργανα που με ρωτήσατε νωρίτερα, έχει η Επιτροπή την ευθύνη, το καθήκον, να επαγρυπνεί ως προς την εφαρμογή των οδηγιών. Την ε, οδηγία για το άσυλο και την προστασία των ετούντων πρέπει να μεριμνά για την ορθή τους εφαρμογή. Και απαντώ στην κυρία Αλφανό εν προκειμένου ότι θα πρέπει η Επιτροπή να είναι ο αποδέκτης των ερωτήσεών σας. Η Επιτροπή είναι εκείνη που έχει την ευθύνη των θεμάτων αυτών και όχι το Συμβούλιο. Σημαντικό για μας λοιπόν είναι αυτό το γραφείο υποστήριξης να θεσπίσει μια καλή μέθοδο προστασίας ώστε να προστατεύει πράγματι ε, τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται την προστασία μας. Και το γραφείο αυτό να ε, συνεργάζεται με την Frontex στο βαθμό του δυνατού. Για δε τη Λιβύη, σε πολιτικό επίπεδο θα σας απαντήσω, δεν είχαμε επαφές. σε ε, ένα πολύ ευρύ πλαίσιο έχουμε αναπτύξει τις επαφές μας με τη Λιβύη και τα θέματα αυτά του ασύλου είναι μόνο ένα κομμάτι των συζητήσεων και των διπραγματεύσεων που έχουμε τη χώρα αυτή. Έχουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων προς συζήτηση. Δυστυχώς όμως υπό τη Σουηδική Προεδρία κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία λόγω της καθυστέρησης που σημείωσαν οι ε, αρχές της Λιβύης ε, ως προς την ανταπόκριση στα θέματα μας και μάλιστα ε, σήμανα και νωρίτερα ότι ταυτόχρονα όταν έπρεπε να επισκεφθούμε τη χώρα ήταν ασθενής, ασθένησε και ο υπουργό αλλά α μην περιοριστώ μόνο στην Λιβύη. Μιλήσατε για την Τουρκία. Είναι μια χώρα με την οποία πρέπει να συνεχίσουμε τι συζητήσει έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα πιο πλήρε με καλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε την επόμενη σειρά ερωτήσεων. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Μια πολιτική συμφωνία όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα εγκατάσταση ε, για την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεσμευτούν και οι 27. Ή θελούσαν να προσχωρήσουν επομένω ε, σε αυτήν την κίνηση τα κράτη-μέλη. Έτσι δεν είναι, κάτι άλλο. Σα είπε ο κύριο ε, Μπούσουτελ ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να αναθεωρήσουμε το καθώς που διέπει την Eurodac και την συνθήκη του Δουβλίνου. Πρόσφατα δε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να κάνει μια αναθεώρηση της ε, ε, απόφασης της οδηγίας για το άσυλο Επομένω, ε, θα πρέπει να αλλάξει τώρα η σημαντική στήλη τη δέσμη ε, μέτρων σχετικών. Για το δικαίωμα στο άσυλο ή για τις προϋποθέσεις προσχωρήσης ασύλου. Ποιο από τα δύο θα πρέπει να αλλάξουμε. Αφού λοιπόν επισημανθεί ποιο είναι το θεμέλιο αυτής της ε, πολιτικής. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει κάποιες προτάσει και θα πρέπει κάτι να κάνουμε πριν το 2012. Προ το παρόν δεν κάνουμε τίποτα. Πετε μου πώ βλέπετε τα πράγματα εσείς. Ο κύριο Μπόντο. Έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει, κύριε Υπουργέ, ο κύριο Μπόντο. Η πρώτη. Ε, κάτι που αφορά την ε, νόμιμη μετανάστευση. Μα είπατε ότι εσεί θέλετε οι στόχοι τη πολιτική Λισαβόνα να συνεχίσουν να ισχύουν, δηλαδή ότι να ε, δεχόμεθα τους αναγκαίους μετανάστες. Μετά όμως ε, δεν μας είπατε κάποιο είδου πιστικά επιχειρήματα γιατί τι θα γίνει με όλες αυτές τις χιλιάδες των ανέργων. Όλοι αυτοί θα συμφωνήσουν μαζί σα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αναδεχόμεθα μετανάστες. Πρώτον. Δεύτερον, μας είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη. Τι εννοείται με αυτό, τι εννοείται αλληλεγγύη. Τι θα γίνει με στα σύνορα, τι θα γίνει με στον οδό αυτή, πρόκειται να ενισχυθούν οικονομικά, διότι θα πρέπει να συνεισφέρουν στην προστασία των σύνορων. Πώς θα γίνει η απορρόφηση των μεταναστών, Πώς θα γίνει η κατανομή επίσης του βάρους αυτής της ζωής μεταναστών. Τι εννοείται επομένως ακριβώς να λέτε αλληλεγγύη. Επόμενος. Κύριε που μα είπατε, λέει ο κύριο Μπρόν, ότι αν γίνει σωστή διαχείριση μεταναστών θα ωφελεί στους πάντες. Για πετε μας όμως, τι θα πούν αυτοί που δεν έχουν δουλειά στα κράτη-μέλη όταν δουν να καλοδεχόμαστε νέου μεταναστές που θα έρθουν να δουλέψουν. Ή έστω αυτοί που έρχονται τούντες άσυλο. Είναι γενεδορία, είναι καλή διάθεση, όμως από την άλλη μεριά η γενεδορία προϋποθέτει θυσία, θυσία αυτού που ερχονται τούντε ασυλο ειναι γενεδορια ειναι καλη διαθεση ομως απο την αλλη μερια η γενεδορια προυποθετει θυσια θυσια αυτου που ειναι ο γενναιόδωρος. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη, και εμείς και εσείς. Αυτοί που θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι θα είναι οι μη προνομιούχοι στα κράτη-μέλη. Ούτε καν θα ωφεληθούν οι χώρες ε, προέλευσης. Έχω εγώ στο χωριό μου κάποιους ε, ε, υπάλληλου του χώρου της υγείας που τους εκπαιδεύουμε και δουλεύουν εκεί πέρα στο χωριό μου. Όμως αυτοί χρειαζόταν να δουλέψουν στο δικό τους χωριό, στη χώρα τους. Σιγά σιγά δημιουργούμε λοιπόν ένα προλαταριάτο. Παγκόσμιο. Παγκοσμιοποιημένο. Γυρούνται σε άσυλο με το που γίνεται δεκτή αίτησή του, σταματάνε να είναι. άσυλο. Γίνονται οικονομικοί μετανάστε. Σε κάποιε χώρε χρειάζεται μετανάστευση, σύμφωνοι και είναι καλοδεχούμενοι όμω. Έχουμε, έχουμε, είμαστε κάργα από του μετανάστε. Δεν χωράνε άλλοι. Δεν μπορούμε να αναδεχθούμε περισσότερου. Eh. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ρίξουμε αυτό που είπε η κυρία Πλάσχαρτ. Σε σχέση με την ε, εγκατάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη, θα είμαι σύντομο γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο θα το συνεχίσει η Ισπανική Προεδρία και η οποία και φυσικά θα συνεχίσει το συζητά μαζί σας. Όπως προείπα θα είμαι σύντομος. Και ήθελα να πω στον κύριο Μπόντε ότι η οικονομική μετανάστευση που μας απασχόλησε στη συνάντησή μα στο Ασβούργο. Ακούσατε και τις απόψεις μου και βέβαια θεωρώ ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ ετούντες άσυλο και μεταξύ εκείνων που είναι θύματα των δουλεμπόρων μεταναστών. Βεβαίω και χρειαζόμαστε την μετανάστευση για να προοδεύσουμε σε κάποιους οικονομικούς τομεί και γι' αυτό και στο πρόγραμμα Στοχόλμης υπάρχει για την νόμιμη μετανάστευση ένα κεφάλαιο, κεφάλαιο που καλύπτει πάρα πολλά θέματα. διαταμένο. Είναι θέμα αυτό του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Σουηδικής Προεδρίας. Τώρα για τις ευθύνες μας όσον αφορά την ε, αλληλεγγύη πρέπει να επιδείξουμε. Έχουμε ξεκαθαρίσει τι εννοούμε, επανειλημμένα. Είπαμε τι σημαίνει αυτό το σύστημα εγκατάστασης που θέλουμε να ε, λειτουργήσει. Οι κάτω χώρες είναι πάρα πολύ προχωρημένες σε αυτόν τον τομέα, όμως θα χρειαστεί ισορροπία μεταξύ των μεθοριακών ελέγχων και από την άλλη μεριά της αλληλοβοήθειας της επίδειξης αλληλεγγύης του ενός προς τον άλλο. Αλληλεγγύη προς κάποιες χώρες που έχουν πάρα πολλούς πρόσφυγες. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με εξισορρόπηση επομένω των επιμέρους θεμάτων και εν ώψη των εξελίξεων της αύξησης των, ε, των που θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Ναι, το περιοδικό πρόγραμμα που αφορά τη Μάλτα, όπω είπατε για μα, είναι ένα μπούσουλα, είναι ένα προπομπό και θα πρέπει να δούμε τι σημασία έχει η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα χωρί μετανάστευση θα ήμασταν φτωχότεροι, θα ήμασταν λιγότερο οικονομικά δυναμικοί. Θα ήμασταν λιγότερο καλοί να αντιμετωπίσουμε τι διάφορε προκλήσει. Οικονομικέ και άλλες. Τα είπαμε στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης Πώς αντιμετωπίζουμε, πώς βλέπουμε την διαχείριση της ε, οικονομικής μετανάστευσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ανάγκε του κάθε κράτου μέλου που φυσικά διαφέρουν από το ένα στο άλλο. Βεβαίω και έχουμε ε, κάποια μέρη και στη Σουηδία που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ας πούμε έχει πάει προσωπικό νοσοκομιακό στη Βόρεια Σουηδία και άρα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και να μην έχουμε κρατικές ιδέες ότι δηλαδή θα πρέπει να μην αφήνουμε ας πούμε νοσοκόμους, νοσοκόμες από την Αφρική να πηγαίνουν αλλού, γιατί πηγαίνοντας αλλού πιάνουν αλλού τη δουλειά, βγάζουν χρήματα, τα στέλνουν στο χωριό τους και έτσι συντηρούν την οικογένειά τους στη χώρα προέλευσης. Δεν θέλουμε να το δούμε σαν νεοαπικιοκρατικό καθεστώς αυτό. Άρα... Δεν θέλουμε να το πάμε εκεί, δεν θέλουμε εκεί να οδηγήσει το πρόγραμμα Στοκχόλμης. Θέλουμε να προσέξουμε το θετικό κομμάτι, δηλαδή πού μπορεί να βοηθήσει η μετανάστευση της ε, χώρες και προέλευσης και προορισμού. Νομίζουμε ότι είναι ένα ρεαλιστικό όραμα και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστούμε κύριε Μπίλστρομ που ήρθατε και μας είπατε όλα αυτά και απαντήσατε αυτές τις ερωτήσεις. για συνεργασία σας. Ε, συγχαρητήρια για τα όσα έχετε καταφέρει και καλή επιτυχία στο μέλλον. Ελπίζουμε δε να τα ξαναπούμε. Eh, Σα ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών για την συνεργασία. Σας εύχομαι πολύ καλά Χριστούγεννα και στο επανειδήν. colleagues, we continue Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα, έχουμε την ψηφοφορία, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ε, εγκρίνουμε τα πρακτικά τις τελευταίες μας συνεδρίασεις Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίας 16 της 10 της 22ης Ιουλίου, 19 Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 2009. Εφόσον δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, προχωρώ στις ψηφοφορίες περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που σχετίζονται με τον Οσάμα Μπιν το δίκτυο της Αλκάιντα και τους Ταλιμπάν. Σε σχέση με τη Ζιμπάμπουε και ε, στρεφόμενα κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων οντοτήτων και συγκεκριμένων οργάνων ενώπιση κατάσταση κατάστασης της Σομαλίας. Πριν από την ψηφοφορία θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπράτλεϊ. Ο πρόεδρος ε, απέστειλε επιστολή και στα μέλη της Επιτροπής μας και στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου ζητώντας πληροφορίες για, τις, ε, για τους τρεις φακέλους που είναι αντικείμενο του ψηφίσματος υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το ζήτημα της νομικής βάσης ήδη συστήθηκε στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Bradley για να μας εξηγήσει αυτές τις πτυχές. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από μερικά χρόνια μια εκπομπή στην ε, Βρετανική τηλεόραση με τον τίτλο «Η ζωή στον Άρη» μιλούσε για έναν αστυνομικό ο οποίος ε, ε, έπεσε σε λίθαργο το 36 και ξύπνησε το 70 κάτι και ε, δεν είχε ακούσει ποτέ του για αυτοκίνητα, δεν είχε ακούσει ποτέ του για γυναίκα πρόεδρο ή πρωθυπουργό κτλ. Όλα αυτά ήταν σαν να μιλάμε για ζωή πάνω στον Άρη, για Αριανούς. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε, στα οποία θα μπορούσαμε να δούμε παραλληλισμούς ως προς τις ε, πεπαλαιωμένες και απειρχαιωμένες προτάσεις, όπως το να φορούσαμε παντελόνια ε, καμπάνα και να είχαμε τα μαλλιά σε στυλ άφρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη νομική βάση 15.2. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους ε, δεν μπορεί να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή επί τη βάση του 215 ε, γιατί βέβαια αυτό αποτελεί οπισθοδρόμηση σχέση με τις ε, εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Το ζήτημα, η ταυτότητα του προτείνοντος οργάνου και η ουσία των προτάσεων που έρχονται από τις Επιτροπές σας. Καταρχάς, τα μέτρα μπορούν να στηριχθούν μόνο στο άρθρο 215 εφόσον ληφθεί απόφαση υπό τον τίτλο 5 άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρώτα απ' όλα χρειάζεται κοινή πολιτική ε, η απόφαση επί της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας του Συμβουλίου. Και μετά, βάσει αυτή, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 215. Εφόσον λοιπόν δεν έχει τηρηθεί αυτός ο πρώτος όρος, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 215. Ως προς την Ζιμπάμπουε, Υπάρχει κοινή θέση βάση του τίτλου 5 αλλά τη συνθήκη πριν από τη Λισαβόνα. Πράγμα το οποίο δεν ταυτίζεται πιστεύω με την, ε, πιστεύουμε με την ε, διάταξη του άρθρου 2 του 5ου τίτλου. Είναι διαφορετική διαδικασία, διαφορετική συνθήκη, διαφορετικά τα όργανα που παρεμβαίνουν στη διαδικασία αυτή και διαφορετική στόχη που εξυπηρετεί, καθώς και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται και όσον αφορά την ΚΕΠΑ και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Κατά την άποψή μας λοιπόν Πρόεδρε δεν είναι δυνατόν να ε, συγκριθεί μια κοινή θέση της ε, πρόλης λισαβονος νομοθεσίας με, την, ε, με το τίτλο, το δεύτερο άρθρο της Λισαβόνας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι επιπλέον για τους οποίους δεν μπορεί η Επιτροπή να προτείνει αυτό το άρθρο. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δράσει μόνο επί τη βάση κοινή προτάσεως του είπα του εκπροσώπου των Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι προτάσει αυτές η Επιτροπή τι υποβάλλει μόνη τη αυτοδυνάμως και κατά την άποψή μα δεν μπορεί ε, διαδικαστικά να είναι ορθή διαδικασία προτείνεται. Επίσης δεν μπορεί το 215 για λόγους ουσίας, για λόγους περιεχομένου των προτάσεων να εφαρμοστεί. Και γιατί περιέχει, για τα θέματα που περιέχει, αλλά και για τα θέματα που παραλείπτει στο 215.3 ως προς παραλήψεις αναφέρεται ότι θα πρέπει να διατίθενται, να αναφέρονται στην πρόταση οι ε, διατάξεις και οι διασφαλιστικές δικλίδες, πράγμα το οποίο έχει ήδη στο παρελθόν προκαλέσει αρκετές δυσκολίες και αντιπαραθέσεις. Εκ των τριών προτάσεων, μόνο η πρόταση για την Αλκάιτα δίνει αρκετά στοιχεία, ενώ οι άλλες δύο παραπέμπουν το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα το οποίο για μας δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 215. Από την άλλη, ε, για τις προτάσεις που αφορούν την Αλκάντα και τη Σομαλία, γίνεται λόγος, γίνεται παραπομπή στην ε, επιτροπολογία 19-19, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει πλέον, διότι γίνεται εφαρμογή, ισχύει η εφαρμογή του άρθρου 202 της, ε, μάλλον αποτελεί εφαρμογή του άρθρου 202 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει καταργηθεί εντωμεταξύ. Άρα μόνο ε, επί τη βάση του δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη. Ας πάμε τώρα να δούμε το, ε, το άρθρο 75 τη συνθήκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του περιεχομένου των μέτρων που προβάλλονται, Αναφέρεται ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, αποφασίζουν ένα πλαίσιο διοικητικών μέτρων όσον αφορά τις, τις κεφαλαίων διαφορών ατόμων ή οργανώσεων. Και πρόεδρε, προσπαθήσαμε να διανοηθούμε τι μπορεί να είναι πλαίσιο διοικητικών μέτρων, γιατί πρόκειται για νέα διαδικασία. Εάν λοιπόν διοικητικά μέτρα είναι αυτά τα οποία προσδιορίζουν το ποιο άτομο και ποια οργάνωση στοχεύονται για το πάγωμα των, των πόρων, τότε δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο βασικούς κανόνες. Άρα θα πρέπει να προσοριστούν και τα, οι πόροι ποιοι είναι και οι οικονομικοί πόροι είναι, ποιοι είναι και το πάγωμα ποιο είναι και το πεδίο εφαρμογής αυτού του παγώματος και η απαγόρευση για οποιαδήποτε συμπληρωματική δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεάσει το πάγωμα και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις διατάξεις περί ε, ευθύνης ε, εφαρμοστικών μέτρων ανταλλαγής ε, πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και επιτροπής και ούτω καθεξής. Το άρθρο 75 έχει περιορισμένο πεδίο ως προς τους στόχους, είναι περιορισμένος προς τους στόχους που μπορεί να επιδιώκονται από κάποιο μέτρο που εισάγονται δυνάμει του. Περιορίζεται δηλαδή σε στόχους καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των συναφών δραστηριοτήτων. Κατά την άποψή μας οι προτάσεις αυτές 2097 θα μπορούσαν να υπαχθούν στα προσαρμοστικά μέτρα του 75 με βάση τον κανονισμό του 2002 και εάν το δούμε τον κανονισμό αυτό, 881 του 2002, στόχος του είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και δεν αλλάζει τίποτα ως προς τη διατύπωση της πρότασης. Το ακολουθεί δηλαδή αυτό η πρόταση. Ως προς το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιείται ο κανονισμός αλλά δεν μεταβάλλεται η ουσία, του, ο χαρακτήρας του ως μέτρο εφαρμοστικό. Δηλαδή παραμένει εφαρμοστική η πρόταση. Πλην όμω θα πρόκειται για νομοθετικό μέτρο εφόσον προχωρήσει με αυτή τη διαδικασία και άρα θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι 8 εβδομάδε για την επαλήθευση τη επικουρικότητα ε, ε, στα εθνικά κοινοβούλια για τι προτάσει αυτέ. Αλλά ούτε για τη Ζιμπάμπουε ούτε για τη Σομαλία φαίνεται να επιδιώκονται οι στόχοι ε, τη καταπολέμηση τρομοκρατία. Γιατί η πρόταση για τη Ζιμπάμπουε μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό του κράτου δικαίου, ενώ τη Σομαλία αναφέρεται σε άτομα και οργανώσεις μάλλον της, της ε, Σομαλίας, ναι, που α, μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη δημόσια τάξη. Άρα, κατά την άποψή μα, δεν είναι δυνατόν κατά την άποψή μα να στηριχθούν αυτέ οι δύο προτάσει, Σομαλία-Ζιμπάμπουε, στο άρθρο 352 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντικατέστη το άρθρο 308, που όπω γνωρίζετε ήταν η γενική ρήτρα. Η ρήτρα πασπαρτού, όπω λέγαμε παλιά, δηλαδή αυτή που εφαρμοζόταν όταν καμιά άλλη δεν ε, έκανε τη δουλειά που θέλουμε. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα του 252 εξασφαλίζεται μόνο εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα για δράση από κάποιο άλλο άρθρο. Για μας υπάρχει δυνατότητα δράσης διαφορετικής είτε από το άρθρο 75 είτε από το άρθρο 215 αλλά στην περίπτωση Συμπάμπουε και της Σομαλίας το Συμβούλιο δεν έχει ασκήσει τις εξουσίες που του προσφέρουν τα εν λόγω άρθρα. Πολύ σύντομα για να απαντήσω στις παρατηρήσεις ε, από την, επιστολή του κ. Λόπερ Σαφίρα δεν μπορούμε να εναλλάξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε υπαλλακτικά τις δύο αυτές ε, διατάξεις, γιατί ή ο ένας στόχος υπάρχει ή ο άλλος. Την ιδέα επιλογή για τις διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο την έχει το Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπορεί να πιέσει, δεν μπορεί να επιβάλλει τις ε, αναλύσεις αυτές στο Συμβούλιο. Πρόεδρε, αυτές ήταν οι αναλύσεις της νομικής υπηρεσίας προηγούμενης τρίτης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, ας ψηφίσουμε. Έχουμε νέα τροπολογίες. Πρώτα, ψηφίζουμε. Την πρώτη τροπολογία της κυρίας Μπόσκορτς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές Νομίζω πως πρέπει να μετρήσουμε. Let's check. Will you, will you use uh, your Do you have, do you have your cars here? Έχετε εδώ τις κάρτες σας. Όχι. Ωραία. Θα σας ξαναρωτήσω λοιπόν. Υπέρ. It's adopted. I It's adopted. Okay, it's adopted. Uh, then amendment uh, seven. Τροπολογία 7. Εγκρίθηκε η 6. 7. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα σε ευχαριστώ συνάδελφοι. Δεν ψηφίζουμε για το 6, γιατί όπως ήδη σας είπα στην αρχή της συνεδρίασης και θα αρχίσουμε με την εξέταση του σημείου 7 της ημερήσιας διάταξης. Τη συζήτηση για την μετάβαση από το ΣΥΣ 1 συν στο ΣΥΣ 2. Τροποποίηση της απόφασης και του κανονισμού. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό έγινε την 1η Δεκεμβρίου και ο κύριος Κοέλιο, ο εισηγητής, θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Στη συνέχεια θα ζητήσουμε από την Σουηδική Προεδρία και την Κομισιόν να το σχολιάσουν και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση. Να σημειώσετε ότι αυτή η έκθεση θα επηρεαστεί από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Μια από πρώτε πρώτες τη Κομισιόν βασίστηκε σε μία μόνο σε αυτό δεν ισχύει πλέον, γι' αυτό και καλείται η Κομισιόν να μας πει την άποψή της για τη συνέχιση αυτού του το, τμήματος του πακέτου. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοέλιο όμως. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο. Όντως, όπως είπατε, είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πριν από λίγο καιρό. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα επιχειρήματα που τότε σας ανέπτυξα. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για τις καθυστερήσεις σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν ε, και κυρίως για το σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις, το ΒΙΣ, και ε, κάναμε και προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο. Τελευταία συνεδρίαση του Τζάι ε, αναβλήθηκε η, το κείμενο για το τέλη του χρόνου. Και τελικά αναβλήθηκε εκ νέου για το τέλος του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ε, το αρνητικό αποτέλεσμα αυτής της δοκιμής θα κρίνει το πώς και πότε θα διαπραγματευτούμε τη σύμβαση με την εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για αυτές τις καθυστερήσεις. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να μπορέσει να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, σε σχέση με τις προτάσεις, όπως ε, γνωρίζετε, έχουν υπάρξει προτάσεις σε σχέση με τον κανονισμό. Θα διατηρηθεί με τη νέα νομική βάση. Φαντάζομαι ότι θα είναι το άρθρο 64 της συνθήκης, αλλά κατ' ουσίαν διατηρείται η νομική βάση και θα έχουμε και την πρόταση του τρίτου πυλώνα που θα πρέπει να επανυποβληθεί και ελπίζω πως η Κομισιόν θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερες διευκρινήσεις για αυτό το θέμα. Σε σχέση τώρα με τα θέματα ουσίας, ε, διατηρείται η κατάσταση όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν θέλουμε να δώσουμε λευκό επιταγή στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να οριστεί μία προθεσμία. Δεν δεχόμαστε πρόταση άνευ χρονικής προθεσμίας. Θεωρούμε πως έχουμε συζητήσει ε, για την διαδικασία μετάβασης. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την συναπόφαση και για την νομική βάση και είμαστε υπεύθυνοι ως αρχή επί του προπολογισμού και πρέπει να συνοδεύσουμε, τι, να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία μετάβαση εσείς Φανταζόμαστε ότι κατά τη μετάβαση από το, στο νέο σύστημα θα πρέπει να ενημερωνόμαστε τακτικά και καταλήλως για να μπορέσουμε να δώσουμε θετική γνωμοδότηση. Όποια και θα είναι η τεχνική λύση που θα υιοθετηθεί, θεωρούμε πως όλα τα νομικά μέσα που έχουμε, στη διάθεσή μας, που έχουμε μάλλον εμείς εγκρίνει θα πρέπει να εφαρμοστούν και θα θέλαμε να επενέσουμε τη λύση από το Global Program Management Board που, έκανε, που βρήκε κατά την άποψή μας τη σωστή λύση και μόνο λυπούμεθα που δεν εξευρέθηκε <laughs> νωρίτερα. Εάν αποτύχει το σύστημα SIS-2, επιφυλασσόμεθα ως Κοινοβούλιο να ζητήσουμε από το ελεγκτικό συνέδριο εις βάθος έλεγχο για την υπόθεση. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να ακούσουμε πια και την Κομισιόν και την Προεδρία και τον υπεύθυνο για τις Προεδρίες για τα θέματα Σέγγεν που είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Ε, ε, ο κύριος Άντες που είναι ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για το Σέγγεν, θα πάρει το λόγο. Tack eh, eh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα μόνο να πω από πλευρά της, Προεδρία, από πλευρά της Προεδρίας ότι διαπραγματευόμεθα από αυτού του θέματος από την υποβολή της πρότασης το Σεπτέμβριο. Καταφέραμε να, εξετα... να δούμε την παράγραφο 3 για τα προβλήματα με την νέα πρόταση που θα υποβληθεί με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ είδα το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου, το έχω εξετάσει προσεκτικά και φαίνεται να συμφωνεί με τη συζήτηση που ακούσαμε και στο Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα που ήδη τα ανέφερε ο κ. Σκουέλιο. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη μετάβραση προς μια νέα τεχνική λύση και το Συμβούλιο θα ήθελα να δείτε τη δημιουργία ενός ε, παγκόσμιου, ε, ενός μάλλον γενικού διοικητικού συμβουλίου, πράγμα το οποίο θα αυξήσει, πιστεύουμε, τη δυνατότητα παρακολούθησης από πλευρά των κρατών μελών του προγράμματος αυτού και θα ε, μπορούμε έτσι να επιβλέπουμε και την ποιότητα. Η συζήτηση τώρα στο Συμβούλιο, βασικά είναι ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν πως είναι σημαντικό να υπάρχει μια τελική προθεσμία και επίσης είδαμε από την, το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θα μπορούσα να σας αναφέρω. Αυτές πιστεύω ότι αφορούν το σχέδιο του Κοινοβουλίου. Συμπεριλαμβάνονται εδώ πτυχές ε, για την λήψη αποφάσεων ε, κατά τη διάρκεια της φάσης ε, μετάβασης από το τωρινό σύστημα δηλαδή στο νέο. Και από ό,τι φαίνεται, με την ισχύουσα νομοθεσία, η Κομισιόν θα πρέπει να έχει καλύτερες, περισσότερες δυνατότητες για να ε, παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Annars så Όπως σας είπα, έχουμε κάποιες κοινέ ιδέες με το Κοινοβούλιο. Έχουμε παρόμοιες ιδέες για το πώς ε, θα μπορούσε να εξελιχθεί η πρόταση της Κομισιόν, ώστε να ε, προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να υιοθετήσει το Συμβούλιο σε σχέση με τη σημασία του Γενικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου. σημειώνουμε τη σημασία της ε, διατήρησης της λειτουργίας του συστήματος μέχρι την εξέβρεση εναλλακτική λύσης και αυτό με οδηγεί και σε κάτι που ανέφερε ο κ. Κοέλιο. Ότι δηλαδή τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Συμβούλιο τη Δευτέρα για το ΣΥΣ αναφέρουν, όπως είπε και ο κύριος Κουέλη, ότι οι καθυστερήσεις που είχαμε μέχρι στιγμής σε αυτό το πρόγραμμα στις δύο δεν μπορεί να συνεχίζονται. Το συμπεράσματα λοιπόν του Συμβουλίου λένε ότι αν δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την τελική φάση των δοκιμών όπως έχει προγραμματιστεί αρχικά για το τελευταίο τρίμηνο του 2004, λέει ο μιλητής, δέχτηκε το Συμβούλιο την παράταση μέχρι τις αρχές του 2010. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Οπότε τότε το Συμβούλιο θα θεωρήσει πως οι δοκιμές αυτές έχουν αποτύχει. Χρειάζεται να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εναλλακτικά τεχνικά σενάρια Και προχωράμε μετά και στην έκθεση του Κοινοβουλίου που λέει ότι η εναλλακτική λύση θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα. ώστε να έχουμε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που περιγράφονται στα νομικά μέσα στο συς Αυτά από το 2006 είναι οι προδιαγραφές να μπορέσουμε να δώσουμε δηλαδή στους πολίτες και στις αρχές πρόσβαση στο ίδιο σύστημα. Θεωρούμε πως αυτό είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Δεν θα σας πω τίποτα σχετικά με αυτό. Αλλά να σας πω πως δεν έχουμε προγραμματίσει άλλες ε, συναντήσεις αυτής της ομάδας εργασίας. Δεν προβλέπονται άλλες κατά τη διάρκεια της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Θα ενημερώσουμε την επερχόμενη Προεδρία πολύ προσεκτικά σε σχέση με τις θέσεις ε, του Κοινοβουλίου. Και θα διασφαλίσουμε την διαρκή ενημέρωση του Κοινοβουλίου για το θέμα και για το τεχνικό επίπεδο του συς Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Πρόεδρος, ευχαριστούμε, κύριε. Και τώρα να ακούσουμε τις απόψεις των μελών της Επιτροπής. Ε, παρακαλώ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, τι έχει να μας πει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επισέλθω στις ε, λεπτομέρειες και στους στόχους της ε, πρωτοβουλίας αυτής και της τροπολογίας, γιατί τα είπαμε την περσμένη εβδομάδα. Όμως, να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις του κ. Κόελιο. <clears throat> Τονίσαμε για τα τεχνικά θέματα, στην τεχνικές λεπτομέρειες, ότι προσπαθούμε να με διαφάνεια, ευθύτητα και στο τεχνοκρατικό τεχνικό επίπεδο. Είχαμε πλευράς ε, σύμβαση κάποια προβλήματα τα είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου νομίζω. Και όλα αυτά τα ζητήματα απαντήθηκαν στην από την γραπτήρα του κ. Κοέλιο κατά την ίδια Ολομέλεια. Πάρα πολύ επικοδομητικό το πνεύμα του κυρίου Κοέλιο, πάρα πολύ επικοδομητικό το κείμενό του. Οι προτάσεις αυτές νομίζω ότι συνάδουν προς το συμβαστικό αυτό κείμενο. Τα είπαμε για το κεκτημένο του Σέγγεν τους ε, τελευταίους μήνες. Αλλά να σας πω τώρα για τα πιο σημαντικά σημεία της έκθεσης. Μερομηνία. Εμείς δεν μνημονεύουμε συγκεκριμένη ημερομηνία με κανένα λόγο για να αποκρύψουμε κάτι, να θολώσουμε τα νερά από το Κοινοβούλιο, για να υπερβάλλουμε όσον αφορά τις τεχνικές ε, δυσκολίες. Απλώς, στη σημερινή συγκυρία δεν ήμασταν σίγουροι κατά πόσον μια τέτοια, ένα τέτοιο πλαίσιο για το ΣΥΣ2 θα ήταν ότι το καλύτερο για να μπορέσει να τρέξει όπως πρέπει. Δεν μπορούσαμε να βρούμε δηλαδή κάποια ρεαλιστική ημερομηνία γιατί η ημερομηνία θα πρέπει να εξαρτηθεί από κάποια στάθμιση και επιλογή από τα σενάρια που είχαν προταθεί. Παρ' όλα αυτά, τα συζητήσαμε όσον αφορά το κείμενο του Σέγγεν και λάβαμε υπόψη το κείμενο Κοέλιο, την έκθεση Κοέλιο. Φυσικά και πρέπει να βρεθεί μια σχετική ημερομηνία τελικά και θα πρέπει όμως να αποφασιστεί κάτι και να επιλεγεί μια λύση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η πλατφόρμα για το ΣΥΣ2 πάει για το τελευταίο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Ε, αναφέρεται και κάτι σχετικά από την ε, έκθεση. Για το ΣΥΣΕΝΑ, 1 συν τώρα είπαμε ότι το 2012 θα μπορούσε να είναι η εναρκτήρια ημερομηνία. Όμω είπαμε ότι μπορεί αυτό να είναι για το 2013. Ακριβώ επειδή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι σήμερα, θεωρήσαμε ήταν ανέφικτο να καταλήξουμε σε μια ημερομηνία την οποία σα προτείνουμε ή ότι μπορούμε να κάνουμε μια τροποποίηση του κειμένου πριν έρθει η ώρα. Πάντω και προκειμένου μα καλύπτει το κείμενο του Σέγγεν, είναι κάτι που ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο και εμεί θέλουμε υποδομητικά να συνεργαστούμε για να βρούμε την καλύτερη λύση και την πιο δόκιμη, πιο κατάλληλη ημερομηνία. Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την ε, ορολογία, τη διατύπωση αυτή τη ίδια τη τροπολογία σε ίση με το ΣΥΣ2. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα το ΣΥΣ2, είπαμε ότι ε, είναι μια νομική ομπρέλα, είναι ένα σύνολο κανόνων και θα μπορούσαμε να βρούμε μια τεχνική λύση για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Επίσης, τα είπαμε αυτά, τα λέει και ο κύριος Κόλλιο, μας ε, χαιροποιεί πάρα πολύ το, ε, η σύγκληση αυτών των απόψεων. Οπότε, για τους ίδιους λόγους η φρασιολογία, η διατύπωση στην έκθεση αλλά και στην πρότασή μας μπορεί να προξενήσει κάποια σύγχυση γιατί περιγράφεται κάποια συγκεκριμένη επιλογή και λύση, ας πούμε, που τώρα κυριαρχεί. Όμως, εμείς νομίζουμε ότι το ΣΥΣ2 θα πρέπει να αναζητηθεί, να καλυφθεί από μια τελική νομική λύση πλαίσιο και έτσι να, να, να, να επιλαγεί κάποια στιγμή μια άλλη πλατφόρμα. Πάντως ε, νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να αναζητήσουμε κάποια λύση εμείς και ο συγητής. Τελευταίο τώρα όσον αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την ε, υπόθεση, για αυτή την πολιτική της μετανάστευσης για αυτή την ε, αλλαγή μεταξύ του ΣΥΣ 1 ε, συν και του ΣΥΣ 2 όταν είναι βέβαια τεχνικά άρτιο το ΣΥΣ 2 και μπορεί να γίνει η μετανάστευση αυτή η μετάβαση. δηλαδή θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει κάποιο ρόλο σε αυτή την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μας, συνάδει προς ε, το θεσμικό πλαίσιο εκείνο που θεωρήθηκε ως νομική βάση για το ΣΥΣ2. Νομίζω είναι το άρθρο 55, γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία της μετάβασης θα πρέπει να γίνει με, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες σχετικέ σχετικές αρμοδιότητες, τις δικές μας τις εκτελεστικές, εσείς έχετε τις νομοθετικές, οπότε πρέπει να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα, τι, ποια, ποια συμβατότητα υπάρχει μεταξύ του τι θέλει να κάνει τι, τι, θέλει να πει, τι προτείνει αυτή η έκθεση, ζητά όσον αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην μετάβαση από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2. Πόσο νομοθετικό ρόλο θα τι αποφασιστικό ρόλο μπορεί να λάβει. Α, και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Ότι αυτή η τωρινή πρόταση του πρώτου πυλώνα καλύφθηκε από την ανακοίνωσή μας πέρασμένες εβδομάδες Ισχύει η πρόταση και συνεχίζεται η διαδικασία. Όμως, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Πώς θα γίνει αυτή η ολοκλήρωση. Ακόμα τα συζητάει η νομική υπηρεσία, ο Γενικός Γραμματέας. Μόλις πάντως αποφασίσουμε Βεβαίω και θα σα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Uh, Πρόεδρο. Έχουμε δύο συναντήσει που θέλουν να λάβουν το λόγο. Και κατόπιν να δώσουμε το λόγο, το λόγο ξανά στον κύριο Κοέλιο. Uh, Εγώ είμαι <clears throat> εισηγητής ε, από την ομάδα των σοσιαλιστών δημοκρατών. Συμμερίζομαι την άποψη του κ. Καελιό ως προς τις ε, καθυστερήσεις στη θέση εφαρμογή του συστήματος ΣΥΣ 2. Δεν ε, είναι δυνατό να μην υπάρχει ε, χρονοδιάγραμμα ως προς την θέση εφαρμογή των διατάξεων και πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει διαρκώς να τηρείται ενήμερο για τα αποτελέσματα των ερευνών, τη διαδικασία της επαναδιάρθρωσης και τους όρους της σύμβασης. Δηλαδή κατά πόσο τηρούνται οι όροι της σύμβασης δεν μπορεί να υπάρξει ο οδήποτε έλλειμμα διαφάνειας έναντι του Κοινοβουλίου. Όπως είχα πει και στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, οι στόχοι προστασίας των δεδομένων πρέπει να τηρηθούν ρητά κατά γράμμα. Και οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούν θα πρέπει να είναι οι πιο αποτελεσματικές. τη, μεγάλη, τη μέγιστη ευθύνη τη φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ευθύνη την οποία φέρει και κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αλλά και για τη μετέπειτα περίοδο, όταν θα λειτουργεί πράγματι το σύστημα, είτε είναι αυτό το ΣΥΣ 2 είτε κάποιο άλλο. Και σας ευχαριστώ. Uh, ja, vielen Dank. Also die Kommission sagt, äh, die Angabe eines klaren Datums für die Inbetriebnahme ist nicht möglich. Εγώ θα ήθελα, νέα καθώς είμαι εδώ στην Επιτροπή, να κοιτάξω μια στιγμή την ε, εντολή για την ανάπτυξη του συστήματος, που ήταν ε, ενισχύ μόνο μέχρι το τέλος του 2006. Η μία καθυστέρηση όμως έφερε την άλλη και όταν μου λένε ότι δεν μπορείτε να μου δίνετε σαφή δεδομένα για την λειτουργία κτλ. Εγώ που έχω, δεν έχω τεχνική διαδικασία, τη τεχνική γνώση, θέλω ότι δεν μπορεί να δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα. Διαφορετικά, μόνο λεπτομέρειες θα μπορούσαν να ε, χρειάζονται ρύθμιστη. Αλλά όταν έχει περάσει ο χρόνος ε, επεξεργασίας για το σύστημα και ακόμη δεν ξέρουμε πότε μπορεί να δαθεί σε εφαρμογή, σε λειτουργία, τι να υποθέσουμε στις μεταφορές, παραδείγματι. Εγώ ήμουν για πάρα πολλά χρόνια μέλος ε, στην ε, Επιτροπή των Μεταφορών. Είχαμε το ζήτημα των ε, ηλεκτρονικών της ηλεκτρονικής ανέχνευσιμοτητα φορτίων εκεί, που επίσης χρόνισε για κάποιους λόγους αδιόρατους. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε πάλι με μεγάλε καθυστερήσει, αλλά για ένα σύστημα το οποίο έχει να κάνει με πολύ λεπτά και ευαίσθητα δεδομένα. Ένα σύστημα το οποίο πρέπει να λειτουργεί εξ αρχή από την πρώτη μέρα που θα μπει σε λειτουργία. Και αδιάκοπα, χωρίς κανένα μελανό σημείο. Εδώ τώρα βλέπω ότι δεν ξέρετε, δεν μπορούν καν να μας πούνε πότε θα τεθεί σε λειτουργία. Αυτό σημαίνει για μένα εκβάθρων αμφισβήτηση του κατά πόσο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Και νομίζω ότι και ο συγητής έχει αντίστοιχε ανησυχίες. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή. Ποιο ήταν το αρχικό σας σχέδιο, όταν ξεκινήσατε το, το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό, τι χρονοδιάγραμμα είχατε υπόψη. Μια και πια λόγω της συνθήκη Λισαβόνα μπορούμε να συμμετάσχουμε στην επεξεργασία. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, συγκεκριμένα κάποια στοιχεία ε, και ενδεχομένω άλλα έγγραφα τα οποία θα μα βοηθούσαν να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση. Γιατί βέβαια το ζήτημα, το κρινόμενο εδώ είναι η διαφάνεια και οι συναδέλφοι που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά εδώ και στον καιρό ήδη έχουν διατυπώσει τι παρατηρήσει και τι επιφυλάξει του προ τη διαφάνεια. Γίνεται λόγος για ένα ε, διοικητικό συμβούλιο. Τι σημαίνει διοικητικό συμβούλιο. Έχουν εκπροσώπωση όλα τα κράτη-μέλη σε αυτό. Management Board. Έχει κάποιος μια συγκεκριμένη λειτουργία ή εκπροσώπηση μόνο τυπική ενδεχομένως κάποιων κρατών μελών. Η διαφάνεια διαφυλάσσεται ή η διαφανεια δεν φυλάσσεται. καταρροκωθεί λόγω της ύπαρξης αυτού του συμβουλίου. Είναι πολύ ασαφή τα πράγματα για μένα. Και επίσης Η νομοθεσία για την μετανάστευση, το νομοθέτημα αυτό, ρυθμίζει την ε, νομική κατάσταση της τη μετανάστευση, αλλά ουσιαστικά προσφέρει μια εντολή ε, ανάπτυξης, η οποία ήδη υπάρχει. Εδώ και πολύ καιρό έχει αναλάβει την εντολή το Συμβούλιο. Γιατί λοιπόν δεν λειτουργεί σε τελευταία σε αυτό κοστίζει και πολλά χρήματα αυτή η καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα πρότεινα, θα είχα την ιδέα να ανατεθεί στο ελεγκτικό συνέδριο να επαληθεύσει αυτό το πρόγραμμα. Κάποιο άλλο τον έφερε νωρίτερα, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και έτσι εξασφαλίστηκε και η διαφάνεια. Εγώ έχω έναντι αυτού του ε, προγράμματο, του σχεδίου, μεγάλε αμφιβολίε, δισταγμού και δυσπιστία να εκφράσω. Άρα, ας μας εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει. Ε, δεν μπορούν να αναπτύξουν το σύστημα. Ε, χτυπάνε στα τυφλά, πηγαίνουν στα τυφλά και δεν έχουν βρει το δρόμο τους ακόμα. Υπάρχουν ποινικέ ρήτρε ενδεχομένω από τη μία ανάπτυξη. Τι υπάρχει σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα θέλαμε περισσότερε πληροφορίε από την Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Ζόμερ. Η Επιτροπή, παρακαλώ. Θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσει. Yes, uh, Um, I would uh, try to take them one by one. Um, would you like me to focus on all of the questions? Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να απαντήσω σε ερωτήσεις. Θέλετε να επικεντρωθώ μόνο σε όλες τις τελευταίες, ε, ερωτήσεις τελευταίας ομιλήτρες ή σε ε, ομιλήτρια σε όλες, λέει η σε ολες ε μαλλον σε ολες λεει ο προεδρος Ω προ την ημερομηνία, ίσω ε, δεν ήταν σαφή τα λόγια μου να το διευκρινίσω για άλλη μια φορά για να μην παρεξηγήσετε για μας στην Επιτροπή το θέμα. Δεν ήταν αν ξέρουμε ή αν δεν ξέρουμε ή αν θέλουμε να δώσουμε κάποια ημερομηνία. Δεν υπήρχε ζήτημα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει το σενάριο τεχνικά, υπάρχει ημερομηνία, συνολικό πρόγραμμα, επιχειρησιακό πλάνο. Έως τα τέλη του 2011 πάμε δηλαδή. Πλην όμω και αφού από τον Ιούνιο του 2009 και ύστερα από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο Μετανάστευσης αναπτύχθηκε ένα εναλλακτικό σχέδιο σε επίπεδο συμβουλίου, συμβουλίου ως προς την ανάπτυξη της υφιστάμενης πλατφόρμας σαν εναλλακτική ε, λύση για την επίτευξη του ε, ΣΥΣ2 σε περίπτωση που το τρέχον σύστημα αποτύχει η αβεβαιότητα αυτή, δεν ξέρουμε λέει, τι θα γίνει σε επίπεδο συμβουλίου, δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε ως προς το τέλος του, του προγράμματος. Γιατί αν μείνουμε στο πρόγραμμα που έχουμε τώρα, πάμε για 2011. Εάν όμω αλλάξουμε και πάρουμε την αναλλακτική πρόταση, για την οποία δεν έχουμε επαρκεί πληροφορίες ακόμη, ήταν κάτι το, στο οποίο δεσμεύτηκε η Γαλλία με μια ε, σύμβαση με μια άλλη εταιρεία, η οποία μας έχει δώσει μόνο κάποιε εκτιμήσεις. Αρχικά 2012, τώρα μας έχουν πάει στο 2013. Με αυτή την βεβαιότητα προτιμούμε όταν διατυπώνουμε τροπολογία να μην αναφέρουμε ημερομηνία. Αλλά όπω είπατε, πολύ ευχαριστώ να κοιτάξω πιο επικοδομητικά και με το Συμβούλιο αλλά και με το Κοινοβούλιο ε, το θέμα και να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για μια ε, ημερομηνία συγκεκριμένη για την, διατήρηση του, για την ανάπτυξη μάλλον του κεκτημένου ή μια άλλη ημερομηνία με ενδεχόμενη ανάπτυξη μέσω της ε, παράτασης μάλλον μέσω της επιτροπολογίας όπως αναφέρεται για τη διαφάνεια των ε, δοκιμών του κύριου Έντζο την ερώτηση. Ε, με βάση τη νομική βάση πρέπει αναεξάμεινο να αναφέρουμε, να αναφέρουμε τα αποτελέσματα του συστήματος, πράγμα το οποίο πράττουμε. Επίσης, οποτεδήποτε ε, υπάρξει ένα ορόσημο, είτε σε λήψη αποφάσεων σε επίπεδο συμβουλίου, είτε σε επίπεδο νέας ε, σύμβασης, ε, κάποιες εξελίξεις, που έχουν το χαρακτήρα του ορόσημου, η ε, Επιτροπή ενημερώνει την Πρόεδρο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών, πράγμα το οποίο έγινε και μετά τον Ιούνιο και θα γίνει και τώρα μετά το Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας και όπως είπα χαραπτός υποβάλλουμε διαρκώς ε, πληροφορίες και επιπλέον η προφορική παρέμβαση παρέμβαση του Αντιπροέδρου στο, στην Ολομέλεια στα τέλη Οκτωβρίου. Και στην προφορική λοιπόν παρέμβαση του Αντιπροέδρου αλλά και στις γραπτές απαντήσεις ε, αναφέρουμε και τις ποινικέ ρήτρε άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής εις βάρος του αντισυμβαλωμένου που έχουμε τώρα και τα ποσά που έχουν δεσμευθεί και τα ποσά που έχουν καταβληθεί πράγματι σε πληρωμές. Αυτό λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχουν εξελίξεις ε, σημαντικές, συμβα... συμβατικές ή άλλες, εμείς ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι... Όσο δεν αφορά το, το, το γενικό σχέδιο για το διαχειριστικό συμβούλιο, το JPMB, αυτόν ακριβώς το ρόλο εξυπηρετεί η ύπαρξή του και υπάρχουν τακτικές συνεδριάσεις που παρακολουθούν και κατευθύνουν, δίνουν προσανατολισμούς στο σύστημα. Ό,τι η απόφαση έχει ληφθεί το τελευταίο εξάμεινο από τον Ιούνιο μέχρι τώρα δηλαδή, ε, ως προς την προετοιμασία του πρώτου ορόσημου, Milestone One, έχουν γίνει υπό την καθοδήγηση του Διαχειριστικού Συμβουλίου, το οποίο είχε καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη αυτού του οροσίμου και άλλωστε είχε αποδείξει την αξία του. Και όπως είπα, η οσδήποτε εκ των κυρίων βουλευτών ενδιαφέρεται, έχει βεβαίως τη δυνατότητα να δει το κείμενο της σύμβασης και της απορρέωσης εξελίξεις. Για το ελεγκτικό συνέδριο θα ήθελα να σημειώσω συμπληρωματικά ότι έχει επισκεφθεί την υπηρεσία μας πολλές φορές στο ελεγκτικό συνέδριο για το συγκεκριμένο αυτό σχέδιο. Το προηγούμενο μήνα μόλις, ε, επί τρεις εβδομάδες παρακολούθησαν διάφορες συμβατικές διαδικασίες ε, του σχεδίου αυτού. Φυσικά, είμαστε σε θέση για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή επίσκεψη του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριο Σκέλιο like to. Θα θέλατε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Mike, only... Ε, Πρόεδρε, τρία τελικά σχόλια πρώτον. Σε σχέση με την ευθύνη μας. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις. Το κοινοβούλιο δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτές. Και δεν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση, γι' αυτό και Προτείνω στο Κοινοβούλιο να δώσει τη συνένεσή του για παράταση της εντολής. Ώστε ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο να μπορούν να έχουν δικαιολογία. Επίσης, δεν είναι ευθύνη μας αν κάτι αποτύχει. Κάναμε το νομοθετικό πλαίσιο με πολύ ταχύ ρυθμό. Συμφωνήσαμε στην πρώτη ανάγνωση και πιστεύουμε πως ήταν καλή ιδέα να γίνει και να υπάρξει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο για το γενικό πρόγραμμα, τότε ήταν που ήταν η αρχή, με τη, σύμφωνα με την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, αν η Κομισιόν εξ αρχής είχε επιτρέψει περισσότερο στο Κοινοβούλιο και στα κάτι μέλη να συμμετέχουν, να εμπλακούν, δεν θα ήμασταν σε τόσο δύσκολη κατάσταση, όπως αυτή τη στιγμή. Δεύτερη παρατήρηση. Καταλαβαίνω γιατί λέει η Κομισιόν αν η αρχική τεχνική λύση που είχαν στον προγραμματισμό τους αποτύχει και αυτό θα το γνωρίζουμε στα τέλη του Ιανουαρίου τα αποτελέσματα του πρώτου οροσίμου δεν γνωρίζουν πότε θα υπάρχει η ε, νέα λύση. Και εγώ θέλω να ε, ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν γιατί ειλικρινά μας είπε πρώτον ότι εκείνο πίστευε πως θα είναι το 2012 και τώρα η επιχείρηση η ίδια μιλάει για το 2013 και κανείς δεν ξέρει αν φτάσουμε τον στο Γενάρη και η ίδια εταιρεία μας πήγε το 2014-2015. Κανείς δεν ξέρει λοιπόν και ακριβώς επειδή κανείς δεν ξέρει, θα πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια η κατάσταση η οποία να διαονίζεται πάπυρον. Εφόσον υπάρξει λειτουργική λύση και πρόοδος, θα πρέπει να έχουμε και πάλι διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο με διαφάνεια να μας παρουσιάσουν την κατάσταση. Τελευταία παρατήρηση. Τρίτη και τελευταία. Κυρία Πρόεδρε, αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Εγώ κατανοώ το επιχείρημα σε σχέση με την εμπλοκή του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Δεν θέλω τώρα εγώ να ξανασυντάξω τις συνθήκε και δεν θέλω να προσβάλλω την Κομισιόν και τις αρμοδιότητες της και τις εκτελεστικές της εξουσίες. Όμως θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη για μεγαλύτερη εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Είμαστε υπεύθυνοι για την απόφαση σε σχέση με το νομικό πλαίσιο είμαστε η δημοσιονομική αρχή και υπήρχε Έχουμε συμμετέχει και επενδύσει πολλά σε αυτή τη λύση και έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε γνώση και να συμμετέχουμε στην ε, διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κάρλος. Κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ. Μια ακόμη συμπληρωματική ερώτηση για τον συγγητή. Γιατί να ορίσουμε ως ε, ημερομηνία το 2013 όταν ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή λέει ότι εάν δεν λειτουργεί ω το 2010 τον Ιούλιο, τότε το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι έχει αποτύχει η διαδικασία. Γιατί θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει περιθώριο μέχρι το 2013. Αυτό δεν το εξηγήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αλλά εμείς συζητάμε το 2011 και αν και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το δεύτερο σενάριο, Δεν μπορούμε να ζητήσουμε το 2011 γιατί θα πρέπει να ξαναρχίσουμε, όχι ακριβώς να ξαναρχίσουμε, αλλά γιατί συνεχίζεται η διαδικασία με τα εργαλεία του S1. Αλλά είναι σχεδόν σαν να ξαναρχίζουμε την ίδια διαδικασία. Και νομίζουμε πως το 2013 είναι μια λογική προθεσμία. Κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι το 2013 θα λειτουργήσει θα έχει μάλλον ολοκληρωθεί. Αλλά είναι αυτό που σας είπα και πριν. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ορίσει μια γραμμή και αν δεν έχουν ετοιμαστεί σωστά τα πράγματα μέχρι τότε, και το η Κομισιόν και το Συμβούλιο με το ανώτερο επίπεδο διαφάνειας θα πρέπει να έρθουν εδώ και να ζητήσουν παράταση. Προτείνεται λοιπόν η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών θα πρέπει να είναι 18 Ιανουαρίου για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 4 Φεβρουαρίου 2010. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Ευχαριστώ την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η απαλλαγή. Έχουμε έξι σχέδια γνωμοδότησης που πρέπει να λάβουμε, να εξετάσουμε και να συζητήσουμε. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο την κυρία Γκάντς να αναλάβει την Προεδρία, διότι πρέπει να αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ. Uh, I know that it's quite late, but I think we should... Uh, η καινούργια πρόεδρος λέει, νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε. Uh, King mentioned that our... Όμως, όπως είπε η King Γκάλ, έχουμε τώρα να κάνουμε αυτή την κοινή συζήτηση όσον αφορά την δημοσιονομική αναθεώρηση για το 2008 όσον αφορά τα θεσμικά όργανα. Οπότε, να σας πω, εκ μέρου του κ. που δεν μπορούσατε να τον παραστεί, να σας πω τα εξής. Όπως προαναφέραμε, έχουμε να κάνουμε με, με, με την αφιόρωση του προπολογισμού του 2008. Έχουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αστυνομίας το οποίο πήρε το πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο. Μαθήματα και σεμινάρια οργανώνονται εκεί. Και αυτό το οποίο προτείνεται είναι, όπως και για τις προηγούμενες χρήσεις, πρέπει η σχολή αυτή, αυτό το κολέγιο, να κινηθεί σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύσει αυστηρά τα του προϋπολογισμού του Κολεγίου της Αστυνομίας. Τώρα υπάρχει άλλη μια πρόταση. Αυτή αφορά την Frontex. Η... Το Ελληνικό Συνέδριο είπε πώς θεωρήθηκαν αξιόπιστα τα λογιστικά στοιχεία και οι λογαριασμοί, θεωρήθηκαν σύνομα όλα τα στοιχεία. Όμω, κατά τη χρήση του 2008, αυξήθηκε η προετοιμασία στη Frontex κατά 29 εκατομμύρια ευρώ. 69% και 13 εκατομμύρια των ε, υποχρεώσεων έπρεπε να κυρωθούν γιατί κρίθηκε ότι αυτό το ποσό δεν μπορεί να το, να το, καλύψει η, εν λόγω κοινωτική υπηρεσία. Άρα, οι πιστώσει υποχρεώσεων, όπως και η διαδικασία προσλήψεων, ε, είναι πλάκη. Και θα πρέπει φυσικά να υπάρξει καλύτερη διαχείριση για τις χρήσεις 2009 και 2010. Όσον αφορά τώρα τα τρία, τα τρία άλλα κοινωνικά όργανα, την υπηρεσία για τα φάρμακα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, είπαμε ότι και εδώ δεν υπάρχει αμφισβήτηση της γνωμοδότησης του Ελληνικού Συνεδρίου. Και το ίδιο ισχύει και για την μονάδα της δικαστικής συνεργασίας. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια μέρα θα εξεταστούν οι τροπολογίες. Έχετε παρατηρήσεις? Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρίσταται κανείς. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτό το αστυνομικό κολέγιο, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επαγρυπνεί όσον αφορά τις σχετικές δραστηριότητες και όπως γνωρίζετε ε, άλλαξαν ε, δύο επικεφαλής δύο τμήματων διευθύνσεων για διοίκηση και για πρόγραμμα. Πρόκειται επίσης να υπάρξει και άλλη μια αλλαγή και επίσης έχουμε τρεις υποψηφιότητες για αντικατάσταση ε, του, του διευθυντού ο θα καθήκοντα τον Μάρτιο του 2010 μάλλον. Επομένω. προφανώς τις προποθέσεις ώστε να γίνει κάποια αλλαγή στη λειτουργία αυτή τη υπηρεσία. Ε, ήδη έχει αρχίσει η συνεννόηση για τα θέματα της διαχείρισης των οικονομικών της ε, υπηρεσίας Επομένως σας διαβιώνω ότι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες. Παρακαλώ εσείς. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, συμμερίζομαι τις απόψεις του εισηγητού για το Frontex καταρχάς, ε, γιατί νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το ότι διαρκώ ζητούνται νέα κονδύλια από τη Frontex, ενώ υπάρχουν όλες οι παρεκκλήσεις, παρατυπίες που σημειώνονται διαρκώς για την, ε, από την, σε επίπεδο Frontex. Και επίσης, σημειώνει τις ε, παρατηρήσεις του ε, δικαστηρίου εισηγητής, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και αντί απλώς να καταγράφει αυτές τις παρατηρήσεις, θα έπρεπε να ζητεί, όπως οφείλουμε να κάνουμε ε, ρητά, να προσδιορίσει η υπηρεσία για του χρόνου συγκεκριμένους στόχους και δίκτες ε, επιδόσεων συγκεκριμένους, μετρήσιμους, έτσι ώστε να κρίνουμε την ε, δράση της. Επίσης, όταν διερωτηθήκαμε γιατί δεν έχουμε εκθέσει ως προς την δράση της Europol και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν γιατί έχουμε για τις άλλες υπηρεσίες και δεν έχουμε για την Europol. Και δεύτερον και πιο γενικά, μια και έχω το λόγο για τα θέματα αυτά, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι πολλά από τα έγγραφα τα οποία μας διατίθενται είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά. Ε, παραδείγματι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κοίταξα εγώ, που έχει άμεση επαφή με τον πολίτη και νομίζω ότι αν κανείς είναι επιφορτισμένος με την επαφή με τον πολίτη, θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια στην πολυγλωσία. Πολυγλωσία δεν μπορεί να είναι μόνο μια διαπίστωση κάποιων ε, δεδομένων, πρέπει να μπορούμε να δώσουμε στον πολίτη όλες τις πληροφορίες που μπορεί να του προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση η Πρόεδρος. Ναι, βεβαίως, για τη Frontex έχουμε συζητήσει επί μακρόν τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι θα έχουμε, ελπίζω τουλάχιστον θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, άλλωστε έχουμε και στην έκθεση αξιολόγηση ε, γράψει αυτό, ότι θα πρέπει η Frontex να προσδιορίσει σαφείς ε, και διαφανείς στόχους Για τα κείμενα που αναφέρατε νωρίτερα, η γαλλική έκδοση θα είναι σύντομα έτοιμη για την έκθεση και η προθεσμία για τις τροπολογίες μπορούσε να είναι η 18η Δεκεμβρίου για η ανδήποτε πρόταση τροποποίησης ε, κτλ. Ερωτώ αν υπάρχουν άλλα σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, τότε εάν ε, προσδιορίσουμε λοιπόν, καταγράφουμε την προθεσμία αυτή, 18 Δεκεμβρίου, τελευταία ημέρα της προσεχούς εβδομάδας, λίγο πολύ τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και η προσεχή συνεδρίαση είναι στις 11 Ιανουαρίου και το όντι την πρώτη μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και την παρουσία σας.